Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, dann fangen wir mit dem zweiten Teil. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω όλους στη συνεδρίασή μας. Πάλι έχουμε web streaming, ε, διαβίβαση δηλαδή μέσω του διαδικτύου. Ξεκινάμε σήμερα με το σημείο 13 και τις διαδικασίες για την σταθεροποίηση, για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής ε, Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας αφενός και του κόσμου Αφετέρου, δίνω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή κύριο Άνταμ Σάινφελτ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καλώς ήρθατε όλοι. Όπως γνωρίζετε, έχουμε να συζητήσουμε τον κανονισμό Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το προσδορισμό κοινών ε, βασικών αρχών. Και την επαλήθευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Λειτουργίας της Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κόσμου Παιδίου. Πρόκειται για μια διαδικασία που θα είναι οικία. Έχουμε να κάνουμε με προϊόντα γεωργικά και αλλιευτικά, ή μάλλον που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αλλία ή στη γεωργία, μιλούμε για την ε, δυνατότητα εισαγωγής των προϊόντων αυτών και έχουμε να προσδιορίσουμε κοινούς κανόνες για την διαχείριση των ποσοστώσεων των σχετικών με τα προϊόντα αυτά και τη δυνατότητα επιτήρηση και παρακολούθηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα βλέπετε όλα αυτά στον κορονομισμό. Προβλήματα δεν γύρονται. Αμφισβητήσεις δεν έχουν προβληθεί από κανένα συνάδελφο. Ένα μόνο θα ήθελα να επισημάνω σε μια τροπολογία σχετική με την οντολογική σκέψη υπαριθμών 3 για να υπογραμμίσω το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι πολύ σημαντικός ως προς την εισαγωγή εκτελεστικών διατάξεων είναι μια τροπολογία αυτή που έχει κάνει δεκτή και το Συμβούλιο, εξού και δεν περιμένω καμία δυσκολία στην έγκρισή της. Και νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε την έκθεση. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ακούσουμε τους σκιώδεις ηγητές. Ο κύριος Δάντη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την δουλειά του. Τον προηγούμενο Ιανουάριο, όπω υπενθυμίστηκε, είχε εγκρίνει σε πρώτη ακρόαση τη Συμφωνία σύνδεση και σταθεροποίηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοσμοπεδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου με στόχο την ενίσχυση και την περαιτέρω επέκταση των σχέσεων, χωρί βέβαια να... με κάθε μάλλον επιφύλαξη των θέσεων των κρατών μελών σε σχέση με το καθεστώς του κοσμοπεδίου. Ε, κατόπιν της συμφωνίας αυτής λοιπόν το ε, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να εγκρίνουν τον κανονισμό που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουμε ενώπιον μπροστά μας. Έχουμε να κάνουμε ένα file tech, έχουμε στόχο ε, να εγκριθεί σε ταχύτητα τους χρόνους έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι διατάξεις και να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή από το προσοχη Ιανουάριο. Σας υπενθυμίζω ότι αυτή η Συμφωνία σύνδεση και σταθεροποίηση είναι η πρώτη που συνάπτεται μεταξύ Ευρωπαϊκής και και περιλαμβάνει πολύ διατάξεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μιας πορείας ουσιαστικής ενοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προαγωγής των ευρωπαϊκών ε, κανόνων για τον ανταγωνισμό, για τις δημόσιες προμήθειες, την ε, πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία των καταναλωτών, στοιχεία απαραίτητα του προτύπου της εσωτερικής αγοράς που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίσεις εκφράζω την ελπίδα οι πολιτικές συνεργασίες όπως προβλέπονται να αποτελέσουν και κίνητρα και παράγοντες διευκόλυνση της ανάπτυξης στην περιοχή ολόκληρη και να προωθήσουν με τον τρόπο αυτό τη σταθεροποίηση. Ευχαριστώ τον εισηγητή και ελπίζω η έκθεσή του να εγκριθεί με, μεγάλη πλειοψηφία από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλους, εισηγητές, άλλους σκιώδεις εισηγητές παρόντες. Θέλει κάποιος άλλος από τους παρισταμένους συναδέλφους να λάβει το λόγο. Όχι. Λοιπόν, τότε η Επιτροπή. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and uh, thank you very much for the opportunity to, to address. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας απευθύνω το λόγο. Ε, είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη που εξέφρασαν τα μέλη ε, και στηρίζω τα σχόλια του εισηγητή και του σκιώδους εισηγητή. Η Συμφωνία Σταθεροποίησης ε, για το Κωσυφοπαίδιο ξεκίνησε το 2016, πρώτη πρώτου και χωρίς κάτι τέτοιο οι ποσοστώσεις αλληλείας που έχουν ε, συμφωνηθεί ε, στην ε, συμφωνία αυτή δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαμε, μάλλον ορίζουμε, την ταχύτητα με την οποία εξετάσατε το φάκελο Μάλιστα, μία μέρα μόλις πριν ο Επίτροπος Χάνο να μεταβεί στην Πρίστινα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ταχύτητά σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, εισηγητής. E, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια που υπογραμμίζουν ότι το έγγραφο αυτό θα πρέπει να εγκριθεί όσο γίνεται πιο σύντομα και ε, να θυμίσω μόνο μια τυπική πτυχή για όσους είναι σήμερα εδώ. Έχουμε ε, την προθεσμία αποβολής τροπολογιών την 11η 11 η στις 12 το μεσημέρι. Έτσι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. genau, danke schön, Ακριβώς, σας ευχαριστώ πολύ. 11. Νοεμβρίου, όντω στι 12 το μεσημέρι, προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών, 28-29 Νοεμβρίου πάντα, ψηφίζουμε στην Επιτροπή μας. Άρα, έχουμε κλείσει έτσι το σημείο 13 και πάμε στο 14 με ένα νέο πλαίσιο εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκία, δηλαδή εξυγχρονισμός Τελωνιακής Ένωσης. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει την αναγκαιότητα του εξυγχρονισμού της Τελωνιακής Ένωσης με Τουρκία. Και η Επιτροπή έχει αναλάβει δράση για την διατύπωση νέων προτάσεων πιο σύγχρονων ε, για τις σχέσεις Τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία στα εμπορικά θέματα, τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακή Ένωση. αφενό αφετέρου, και το γνωρίζουμε όλοι βεβαίω υπάρχουν μεγάλες πολιτικές προκλήσεις στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Ως εκ τούτου, είναι περισσότερο από απαραίτητο να ε, ξανααναλογιστούμε τις σχέσεις μας και τις εμπορικές με την Τουρκία. Εξού και έχουμε αυτή την έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας με τον κύριο Μπορέλη. Έκθεση η οποία ε, έχει πολύ καλή ποιότητα, ένα πολύ καλό έγγραφο λοιπόν και δίνω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Έχει, θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω, γιατί αυτό είναι το καθήκον μου, τη λογική του στόχου στη δομή του εγγράφου που έχουμε επεξεργαστεί κατά την προετοιμασία του μη νομοθετικού διατάγματος για ένα νέο εμπορικό πλαίσιο και τον εξυγχρονισμό της Θελωνιακής Ένωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Πριν επισέλθω στις λεπτομέρειες, θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση υπό το φως και των πρόσφατων εξελίξεων σε σχέση με τις ισορροπίες, τις ελευθερίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Τουρκία. Δεν μπορούμε εμείς ως βουλευτές να κλείσουμε τα μάτια ενώπιον των πρόσφατων εξελίξεων. Ήθελα λοιπόν να αποτελέσει μια, προ... μια βάση κοινή για συζήτηση το έγγραφο το οποίο σας καταθέσω και ένα πλαίσιο αναλογισμού ως πρώτο βήμα προς τον προσδορισμό μιας κοινή θέσεως. Ε, και βεβαίως οι προτάσεις, οι συμβουλές, οι επικρίσεις που θα διατυπώσετε ενδεχομένως ε, θα αξιοποιηθούν, θα αξιολογηθούν και βέβαια ε, ιδιαίτερα ως προς το εμπορικό σκέλος, αλλά και σαν σύνολο στις δράσεις με βάση τις δράσεις και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Η πρόταση λοιπόν που βλέπετε είναι διαρθρωμένη σε πέντε τμήματα. Έχει υπάρχει καταρχάς ε, ο προσδιορισμός της κατάστασης όπως έχει τώρα, οι πιθανές γραμμές της ε, εξέλιξης, και τα συμπεράσματα με μια εισαγωγή διαπιστώσεων όπου εντοπίζουμε στόχους για να μην ε, χάσουμε τον προσανατολισμό μας σε σχέση με ζητήματα για τα οποία δεν έχουμε με συντολή που όμως μας απασχολούν και είναι ε, υπαρκτά. Έτσι λοιπόν η ε, έκθεση αυτή εγγραφέται σε δύο κατευθυντήριες γραμμές. Καταρχάς την εντολή που έχουμε ως Επιτροπή ΙΝΤΑ, τομεακού δηλαδή χαρακτήρα αρμοδιότητες που δεν μπορούν να επισέλθουν σε ε, άλλα θέματα εμπορικών σχέσεων και δεύτερον μια ευρύτερη προσέγγιση, στρατηγική προσέγγιση που έχει έναντι του υπόλοιπου κόσμου η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια συγκεκριμένη προσέγγιση και σε βάση, με, βάση τις αξίες μας. Ε, στο δικό μας λοιπόν τομέα θέλουμε να ε, συμβάλλουμε στην εξασφάλιση μια προσθέμενης αξίας για τις κοινέ δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τελωνιακή Ένωση, η οποία έχει συμπληρώσει 20 χρόνια, έχει φέρει βέβαια ανάπτυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και για την Τουρκία. Δεύτερον, η γεωγραφική εγκύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από την ε, πρόοδο της παγκοσμιοποίησης και επίσης ανεξαρτήτως τη απόφαση η οποία θα πρέπει να ληφθεί, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτή θα ισχύσει για πολλά χρόνια. Αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη οι συνομιλητές μας και εμείς βεβαίως και ως προς το γενικό πλαίσιο. Υπάρχουν αρκετές ε, σκέψεις, τις οποίες, εκ των οποίων όμως ορισμένες θεωρώ προτεραιότητα. Ε, πρώτον, η Τελωνιακή Ένωση είναι το μόνο διαρθρωτικό κανάλι διεύλος ε, διαρθρωμένου διαλόγου με την Τουρκία που παραμένει ενεργός ακόμη και αυτό Ήδη εχθές ακούσαμε τον ε, πρόεδρο του HDP, του Κουρδικού Κόμματος που ήρθε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξέφρασε πλήρη υποστήριξη και συνένεση ως προς την ενίσχυση των τελειωνιακών εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία ως μόνο τρόπο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η Τουρκία να ε, απομονωθεί. Ε, δεύτερον, ε, η μη εφαρμογή της ε, Συμφωνίας της Άγκυρας, το κομμάτι που αφορά την Κύπρο δηλαδή, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι όρια εκ των για οποιαδήποτε συμφωνία. Σε σχέση με την Τελωνιακή Ένωση και πέραν του δικαιικού πλαισίου έχουμε επισημάνει λοιπόν τα προβλήματα που βλέπουμε και ποιοι είναι οι παράγοντες ε, του τομέα αυτού ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας που έχουμε εντωμεταξύ πολλές φορές ε, ακούσει σε προπαρασκευαστικές επαφές με δύο σημαντικούς τομείς που αναπτύσσονται ως προβληματισμοί Καταρχάς, ε, η ανάπτυξη από πλευράς τουρκικής ε, διαφόρων διαταγμάτων και διατάξεων που εισάγουν ε, τελωνιακούς δασμούς και άρα παραβιάζουν τελωνιακή ένωση και δεύτερον, η ασύμετρη σχέση των τελωνιακών σχέσεων και συμβάσεων που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με τρίτες χώρες και η έλλειψη ε, συνεννόησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυνατότητες για ανάπτυξη των μέλλον συμβάσεων και συμφωνιών ε, δίνει τρία διαφορετικά σενάρια. Πρώτον, τη διαφύλαξη του status quo, δηλαδή τελωνιακή ένωση που ανέρχεται στο 1995 χωρίς καμία τροποποίηση. Δεύτερον, εξυγχρονισμό της τελωνιακής ένωσης για, πιο, για μια πιο ισορροπημένη εξέλιξη ε, όπου θα συμπεριληφθούν και οι αποκλείστατες μέχρι τώρα τομείς και τρίτον αντικατάσταση της Θελωνιακής Ένωσης από μια ελεύθερη και συνολική ε, ε, εμπορική σχέση όπως έχουμε δει να αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια τα σχετικά πρότυπα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει, εάν προχωρήσουμε σε αυτό, να μιλήσουμε και για γεωργία, δημόσιες προμήθειες, υπηρεσίες, ενέργεια, τους τομείς δηλαδή που μέχρι τώρα αποκλείονται από την Τελωνιακή Ένωση τα συμπεράσματα της μελέτης ε, επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στη τελευταία ανάλυση και το πλαίσιο της εντολής μας ε, και η σχετική γνωμοδότηση της ΟΚΕ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη εν προκειμένου. Επίσης, η αξιολόγηση της εντολής μας έχει πολύ μεγάλη σημασία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και τα όρια της θεσμικής μας παρέμβασης ως Επιτροπή ΣΥΝΤΑ, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο δράσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχει μια πραγματική θεσμική αλλά και πολιτική προσθεμένη αξία, θα πρέπει να ε, μπορούμε να στοχεύσουμε σε δύο τύπους αποτελεσμάτων. Πρώτον, συγκεκριμένες, σαφείς προτάσεις για το συγκεκριμένο θέμα της Ελληνικής Ένωσης και δεύτερον, ενίσχυση των κοινωνικών ε, συνδικαλιστικών ε, ε, στοιχείων των δικαίων όπως αυτά αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε τομέα πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ενώπιον μιας σοβαρότατης πρόκλησης, είναι ιστορικές οι στιγμές, αλλά μιας πρόκλησης η οποία θα επιτρέψει να φέρει χρήσιμα αποτελέσματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πάνω απ' όλα για την Τουρκία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος Λάγκη, σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα να δώσω το λόγο στον σκιώδη εισηγητή ο κ. Πάμπριξ του Λαϊκού Κόμματο. Ευχαριστώ πολύ, Μπέρντ. Συμφωνώ με πολλά από τα όσα ανέπτυξε ο κ. Μπορέλη. Το υφιστάμενο πλαίσιο σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ε, ισχύει ήδη από το 1995, δηλαδή κοντεύουμε πια τα 27 χρόνια. Άλλαξαν μεταξύ πολλά πράγματα και αν θέλουμε να κάνουμε πιο επίκαιρους τους οικονομικούς δεσμούς μας και θέλουμε να το κάνουμε αυτό και όχι μόνο, πρέπει να προχωρήσουμε. Βεβαίω υπάρχουν και πολλές παρενέργειες, όμως πρέπει να τηρήσουμε την εντολή μας. Να ανανεώσουμε δηλαδή την τελωνιακή εντολή, που βεβαίω δεν πρόκειται να επιλύσει όλες τις διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Αλλά γενικά, εάν εξετάσουμε την προοπτική, η οδός που έχουμε λάβει ως τώρα βρίσκω ότι είναι σωστή και έχει καλώσει. διότι αυτό άλλωστε απαιτείται και από τους δικούς μας παραγωγούς, εξαγωγής κλπ. και αυτούς που απασχολούνται στις βιομηχανίες αυτές. Αναμένω λοιπόν να υπάρξει σημαντική πρόοδος. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για τα θέματα της Τελωνιακής Ενώσεως το δυνατόν συντομότερο, μη λησμονώντας ότι όπως είπα η προσπάθεια αυτή δεν θα λύσει τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει χρειάζεται μια ενημέρωση, μια επικαιροποίηση ε, στις σχέσεις μας και θα δώσει και μεγαλύτερη, και μεγαλύτερη δυνατότητα άσκησης επιρροής από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα τεκτενόμενα στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Ντάντι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Μπορέλη για το έγγραφο του, το οποίο αποτελεί μια πολύ καλή βάση ε, μελέτης ε, νόψη κυρίως των δυσκολιών των προβληματισμών που αντοπίζουν οι ενδιαφερόμενες πλευρές σε σχέση με την εφαρμογή της τελωνιακής πολιτικής ε, θα πρέπει ταχύτατα να ασχοληθούμε με τις συγκεκριμένες προτάσεις για την ανανέωση του εμπορικού πλαισίου των σχέσεων με την Τουρκία και υπό το φως της προτάσεως και της που θα παρουσιάσει, για την εντολή που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, επιτρέψτε μου, γιατί είναι απαραίτητο αυτό να εντάξω τις, τους πολιτικούς μας στόχους στο υφιστάμενο πολιτικό πλαίσιο. Οι πρόσφατες εξελίξεις Τουρκία ε, προξενούν ιδιαίτερη ιδιαίτερα την προσοχή, προσελκύουν ιδιαίτερα την προσοχή από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και για λόγου γεωγραφικού, όπω γράμισε ο συνάδελφο, η εγκύτητα τη Τουρκία μα υποχρεώνει να ε, παρακολουθούμε, δεν μας επιτρέπει να κλείνουμε τα μάτια στα τεκτενόμενα. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει εκφράσει εδώ και αρκετό καιρό πλέον τη βούλησή της να ε, ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η απόπειρα πραξικοπήματος του προηγούμενου Ιουλίου ήταν ε, ε, μια πράξη κατά της δημοκρατίας, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε αντιδράσεις ε, δυσανάλογες, μαζικούς, μαζικές απολύσεις, φυλακίσεις εις βάρος των μελών της αντιπολίτευσης, το κίνδυνο επαναφοράς της θανατικής ποινής, που απομακρύνουν από το κράτος δικαίου και από τη διαδικασία της ένταξης ταυτόχρονα την Τουρκία όλο και περισσότερο, ήδη έχοντας ε, ως κακό παρελθόν τη μη εφαρμογή του πρωτοκόλου της Άγκυρας για την Κύπρο. Οι αρχές λοιπόν και οι αξίες που μα χαρακτηρίζουν πρέπει να υπογραμμιστούν για άλλη μια φορά και στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση ρητά. Είμαι πεπισμένος εν προκειμένου ότι πρέπει σήμερα να, ε, να αξιοποιηθούν τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ξεκινώντας ακριβώς από αυτά τα εμπορικά μέσα για να ξαναφέρουμε στον ορθό δρόμο το σημαντικό αυτό εταίρο το δρόμο δηλαδή της ε, ενσωμάτωσης, της ένταξης και της σταθεροποίησης, ή της ολοκλήρωσης και της ε, σταθεροποίησης. Οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας παραμένουν πολύ σημαντικές. Το νομικό σύστημα μέσα στο οποίο εγγράφονται είναι βέβαια ξεπερασμένο, το αναγνωρίζουμε αυτό. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε λοιπόν περισσότερο το πώς μπορούν να αρθούν τα εμπόδια που επεσήμανε και ο ομιλητής και τα οποία δεν επιτρέπουν την πλήρη ε, εφαρμογή της Θελωνιακής Ένωσης αυτή τη στιγμή με ένα σύστημα επίλυση διαφορών πρώτα απ' όλα, ένα σύστημα επίλυση διαφορών που θα είναι αποτελεσματικό και που θα κάνει σεβαστό, ε, σεβαστές τις διατάξεις όπως προβλέπονται από τη Συμφωνία για την Τελωνιακή Ένωση και βέβαια η επέκταση των τελωνιακών μας σχέσεων με την Τουρκία στις υπηρεσίες, στις ε, δημόσιες προμήθειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αηφόρο ανάπτυξη και όλα αυτά σημαίνουν πως θα πρέπει ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στο θέμα του σεβασμού και της αμοιβαιότητας των προδιαγραφών, τόσο περιβαλλοντικών, όσο και εργασιακών, όσο και κοινωνικών, όλα αυτά μέσα σε ένα έγγραφο. Και πιστεύω ότι η διάσταση αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία, στρατηγική σημασία. Επί τη ευκαιρία καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για τα πιθανά σενάρια πάνω στα οποία εργάζεται. Ευχαριστώ πολύ ε, τον συνάδελφο και προσβλέπω σε πολύ καλή συνεργασία για το μέλλον. E Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σταρμπάτη. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε με την έκθεση, όπως είπαν και οι άλλοι. Και είναι θαυμάσια η βάση αυτή για την συνεργασία μας. Ο εισηγητής ανέπτυξε τις δυνατότητες για τις μελλοντικέ δράσεις, status quo, εξυγχρονισμός του status quo και οικονομική συμφωνία. Να φύγουμε από το status quo διότι προκύπτουν δυσαρέσκειες και από τις δύο πλευρές. Τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας τα αναπτύξω. Άρα, εξυγχρονισμός της συμφωνίας ή free trade agreement που είναι και το προτιμότερο. διότι αυτό θα οδηγήσει και σε μια απελευθέρωση και στους απομένοντες τομείς. Αυτά θα φανούν από τις διαπραγματεύσεις. Είτε λοιπόν εξυγχρονισμός ή ε, συμφωνία ε, ελευθέρου εμπόριου. Γνωρίζουμε τις εξελίξεις όλοι στην Τουρκία και δεν μας ικανοποιούν, για να το πω πάρα πολύ προσεκτικά. Από την άλλη μεριά λέχθηκε και συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να δούμε, να φροντίσουμε δηλαδή, να παραμείνει κοντά μας η Τουρκία, ασκώντας επιρροή. Εφόσον ούτως ή άλλως σκοτεινιάζει ο ορίζοντας της ένταξης, σωστό είναι τουλάχιστον να προωθούμε τι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Σχάκη, για τους ε, ε, εξονομάτους των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Λέχθηκαν ήδη πολλά. Και βεβαίω έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπω και όλα όσα έχουν σχέση με την Τουρκία, επειδή εγώ είμαι και στην Επιτροπή Εξωτερικών και στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. Θα μιλήσω σήμερα περισσότερο για τα εμπορικά θέματα, αλλά υπάρχουν πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία επίση έχουν προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ενώσεω Τουρκία. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ανάπτυξη του θέματος. Νομίζω ότι βρίσκεται πάνω στη γραμμή με την οποία συμφωνώ και εγώ. Έχουμε μια κατάσταση στην Τουρκία που ε, απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία προετοιμάζει αποστολή για το τέλος του έτους. Όταν πριν από 25 χρόνια αναπτύχθηκε η Τελωνιακή Ένωση είχε θεωρηθεί ως ένα βήμα προς την ένταξη η οποία αναμενόταν πολύ συντομότερα από ό,τι φαίνεται να, γίνει, να μπορεί να γίνει τώρα. Πρόκειται για ένα απειρχιωμένο πλέον πλαίσιο και ο συγχρονισμό του είναι αναγκαίο. Όμω δεν μπορεί να αγνοηθεί και το συνολικότερο πλαίσιο και είναι σωστό να το θέσει ο εισηγητή. Επίσης πρέπει να πούμε σαφώς ότι στη σχέση μας με την Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινείται μόνον από τα συμφέροντα, κάτι που φαίνεται να διαγράφει μια τάση τελευταία. Πρέπει να δούμε βεβαίως τι θα κάνουμε με την επικαιροποίηση της Τελωνιακής Ένωσης. Πρέπει να δούμε και πώς μπορεί να πιεστεί η Τουρκία Πώ μπορούμε να ενισχύσουμε ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνε, σύστημα εμπορίου βασισμένο σε κανόνε και να δούμε πώ μπορούν να συμβαδίσουν χέρι με χέρι αξίε και εμπόριο. Σε ό,τι αφορά τι κρατικέ παρεμβάσει στην τουρκική οικονομία, υπάρχουν πολλοί τομεί που προκαλούν ανησυχίε, Διαφάνεια, αντιμετώπιση τη διαφθοράς, αλλά βεβαίω και στο ψηφιακό εμπόριο. Το ψηφιακό εμπόριο γίνεται όλο και σημαντικότερο. Προσφέρει μεγάλε ευκαιρίε. Επιτρέπει δηλαδή να απολαμβάνουν οι άνθρωποι πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες. Όμως, λογοκρισία ή καμιά φορά και αποκλεισμό ορισμένων ε, ψηφιακών υπηρεσιών ενδέχεται να παρεμποδίσουν σοβαρά την πρόοδο στον τομέα αυτό. Είναι λοιπόν σημαντικό να εξετάσουμε ιδιαίτερα τα πρότυπα και αξίες που θα πρέπει να συμβαδίζουν με οποιαδήποτε πρόοδο της Τελωνιακής Ενώσεως και να εξετάσουμε πώς μπορούμε να εντάξουμε τα υψηλά αυτά πρότυπα, προδιαγραφές στους κανόνες για τη συνεργασία μας με την Τουρκία. Τέλος, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς ό,τι αφορά την εντολή για την επικαιροποίηση, ώστε να μην καταλήξουμε σε μια επανάληψη του θεάτρου εντό εισαγωγικών που είδαμε τελευταία με την πολιτικοποίηση των εντολών και με τη συμμετοχή κοινοβουλίων και άλλων. Να είμαστε σαφείς να έλθουμε σε επαφή και σε συνεργασία με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, stakeholders δηλαδή, και να καταλήξουμε σε μια πραγματική, σε ένα πραγματικό μάλλον εξυγχρονισμό της ε, Τελωνιακής Ενώσεως, χωρίς να κλείσουμε βέβαια τα μάτια μας στους υπόλοιπους παράγοντες. Ευχαριστώ πολύ. Helmut όχι. Η κυρία Σκα Όλοι γνωρίζουμε βέβαια ποια είναι η κατάσταση στην Τουρκία και τις τελευταίες εβδομάδες έχει οξυνθεί ακόμη περισσότερο. Γνωρίζουμε ότι είναι ανύπαρκτη η ελευθεροτυπία. Ολόκληρη την αντιπολίτευση κινδυνεύουν να βάλουν στις φυλακές, ήδη τώρα με το ΧΑΝΤΕΠΕ και με τα εντάλματα συλλήψεως που εκδίδονται για λογαριασμό τους. Θα πρέπει αυτό να έχει κάποιες συνέπειες συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να μην κοπούν όλοι οι δεσμοί και ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί ανοιχτός ο διάλογος. Παρ' όλα αυτά, ο εξυγχρονισμός και διεύρυνση της Τελωνιακής Ενώσεως αποτελεί λάθος μήνυμα για την ώρα. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια αναμένεται νέα συζήτηση για την ε, Τουρκία και οι πιο πολλοί θα πούν τότε ότι οι θεσμοί πρέπει να στείλουν ξεκάθαρα μηνύματα στην Τουρκία. Θα είναι λάθος εάν τώρα εμείς στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου προχωρήσουμε εν σιγή σε εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ενώσεως. Νομίζω ότι στέλνουμε, στέλνουμε το λάθος μήνυμα. Να φροντίσουμε, να ρίξουμε το βάρος μας, να μην προχωρήσουμε τον φάκελο αυτό, να μην ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει εντολή. Πρόκειται για μια από τις λίγες δυνατότητες που έχουμε για να στείλουμε πραγματικά ένα ξεκάθαρο μήνυμα, αν δεν θέλουμε να αποκόψουμε τελείως τους ε, δεσμούς. Άλλοι μιλούν για απόλυτο πάγωμα της ενταξιακής ε, διαδικασίας και διάφορα άλλα. Αλλά πάμε να φτιάξουμε μια, μια τελωνιακή ένωση που είναι και πολύ περισσότερο από μια συμφωνία εμπορίου και να λέμε ότι θέλουμε να την εξυγχρονίσουμε και να την βαθύνουμε, την τελωνιακή ένωση δηλαδή, νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου είναι ε, λάθος μήνυμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μαυρίδης. Thank you, Chairman. I was speaking my mother tongue. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, χαιρετίζω την αναφορά που έχει ήδη ότι στις υποχρεώσεις της Τουρκίας μέσα στην τελωνιακή σύνδεση περιλαμβάνονται και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της είναι υποχρεώσεις δηλαδή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν ένα κράτος μέλος, την Κυπριακή Δημοκρατία, με την οποία αρνείται επίμονα να την εφαρμόσει. Και μπορεί η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι ένα μικρό κράτος μέλος, αλλά είμαστε ισότιμοι Ευρωπαίοι πολίτες και θα υπερασπιζόμαστε οποιονδήποτε Ευρωπαίον πολίτη με το ίδιο σθένος που αναμένουμε να υπερασπιστείτε και εσείς εμάς. Συνεχίζω λοιπόν και θα είμαι πολύ σύντομος με κάποια συγκεκριμένα σημεία. Έχει λεχθεί ότι η τελωνιακή σύνδεση της Τουρκίας ξεκίνησε από το 1994 θα συμφωνήσετε όμως μαζί μου ότι δεν είναι θέμα χρόνου, ούτε έχουμε ευθύνη εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχει εκπληρωθεί. Είναι θέμα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Τουρκίας. Δεν γίνεται να ζητάμε από άλλα κράτη να τηρούν τους κανόνες δικαίου, the rule of law, και εμείς να κλείνουμε τα μάτια θεωρώντας ότι τέτοιες εμπορικές σχέσεις μπορούν να προωθούνται ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις και συγκεκριμένα τις μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και χαρακτηριστικά, όπως πολύ σωστά έχει ήδη αναφερθεί και χαίρομαι γιατί αυξάνονται οι συνετές φωνές. Χθε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υπεθέσεων τέθηκε το ζήτημα για πρώτη φορά για πάγωμα των ενταξιακών της Τουρκίας. Για ποιο λόγο διότι ουσιαστικά δεν εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες δικαίου, δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, υπάρχουν μαζικές παραβιάσεις των θεμελιακών ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων και χαρακτηριστικά την προηγούμενη μέρα ο αρμόδιος επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιέγραψε την κατάσταση με τέτοιο μελανό τρόπο που για να είμαστε αντικειμενικοί πρόκειται για μένα καθεστώς δικτατορίας του Ερτογάν. Υπάρχουν άνθρωποι στην Τουρκία που αναμένουν από εμάς να προασπιστούμε αυτές τις αξίες και είναι απογοητευμένοι. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με μια μόνο επισήμανση. Αφήνω στο περιθώριο την όποια πολιτική συζήτηση ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό για αυτή την αναβάθμιση που συζητάμε των εμπορικών σχέσεων της Τουρκίας. Πέραν από τα πολιτικά, είναι και νομική υποχρέωση. Δηλαδή, εμείς συνεχίζουμε ως να μην συμβαίνει τίποτα και οι νομικές υποχρεώσεις ενός κράτους το οποίο είναι σε ενταξιακό καθεστώς δεν εκπληρώνονται και εμείς θα συζητήσουμε την αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων νομίζω πολύ σωστά έχει λεχθεί και από τον συνάδελφό μου τον κύριο Τάντζη αλλά και από άλλους ότι έφτασε ο καιρός να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και πρωτίστως τα εμπορικά εργαλεία για να ασκήσουμε οικονομικό κόστος πάνω στην Τουρκία. Κλείνω με μια ερώτηση και θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Τηρουμένων των αναλογιών, το τονίζω, τηρουμένων των αναλογιών. Έχουμε ένα αναδιόμενο Χίτλερ. Και ξέρετε σε ποιον αναφέρομαι. Δηλαδή κάποιοι από εδώ θα συζητούσαν την αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων με ένα τέτοιο καθεστώς, ώστε να μην συμβαίνει τίποτα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Ρόισαου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα καταρχά να διευκρινίσω ότι αντικαθιστώ την Μαρίν Λεπέν που δυστυχώ δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα. Ε, πρέπει να μα ρωτήσετε αν θέλουμε να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία ελευθερών συναλλαγών με την Τουρκία. Εγώ πιστεύω πω όχι για δύο βασικού λόγου. Πρώτον, δεν είναι αναπόστατο τμήμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αποκλεί, αποκλίνει όλο και περισσότερο από τι αρχέ μα. Η αυταρχική εξουσία του Ερντογάν διοργάνωσε την απόλυση δεκάδων χιλιάδων ε, δικαστών, αυστυνομικών και υπαλλήλων, κρατικών υπαλλήλων που δεν έχουν καν το δικαίωμα να φύγουν από τη χώρα. Ε, συλλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι ε, και η κουρδική μειονότητα ε, υποφέρει. Εξάλλου παίζει διπλό ρόλο στη Συρία, το γνωρίζετε. Περνά το πετρέλαιο που παράνομα προέρχεται από τη Συρία και, χρηματοδοτείται από, και χρηματοδοτεί έτσι το ΝΤΑΕΣ. Επίσης, βάλει κατά των Κούρδων της Συρίας που είναι ο καλύτερος στρατός που ε, που καταπολεμά του Ισλαμιστέ. Αν κάνουμε τέτοιο είδο λοιπόν εμπορική συμφωνία, θα σήμαινε αυτό κατευθείαν άρνηση των αξιών μα των ίδιων. Έπειτα δεν έχουμε κανένα οικονομικό συμφέρον ε, ούτε στην αγορά ούτε στις εξαγωγές της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν παίζει το ρόλο που πρέπει και ε, σκληραίνει τις, ε, τους ελληνικούς δασμούς. Επίσης δεν θέλει να συμμετέχει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Τέλος, ο ελάχιστος μισθός στην Τουρκία είναι 350 ευρώ Δηλαδή, οι υπαλλήλοι μα ε, μπαίνουν σε ανταγωνισμό με Τούρκου υπαλλήλου που παίρνουν σαφώ χαμηλότερου μισθού και πολλέ επιχειρήσει έχουν μετεγκαταστήσει τα εργοστάσια του. Έχουμε και μάλιστα ένα απόσπασμα της υπηρεσίας ε, αποσχόλησης της Τουρκίας με 20 εκατομμύρια που μπαίνουν στην Τουρκία χάρη στις εξαγωγές. Η χώρα έχει σπάσει το ρεκόρ εξαγωγών το 2015. Δεν πιστεύετε ότι οι ε, εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης έχουν αρκετά υποφέρει από τις χώρες χαμηλού κόστους όλα μας καλούν να μην κάνουμε νέα συμφωνία ελευθερών συναλλαγών με την Τουρκία και δεδομένε της αυταρχικής ε, ε, κλίσης ε, της κυβέρνησης θα πρέπει να σταματήσουμε και τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο σκιώδης συζητητής μας δεν είναι παρόν. Θέλω να πω λίγα λόγια ε, ε, θίγοντας και αυτά που είπε ο κύριος Μαυρίδης. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την ανάλυση των δραματικών γεγονότων στην Τουρκία συμφωνούμε. Είναι απολύτως απαράδεκτα τα όσα συμβαίνουν στην χώρα αυτή αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η διάσταση εμπορικής πολιτικής των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ενίσχυση, αλλά ίσως για την ώρα να μην είναι σωστό να αποφασίσουμε πράγματι. Εγώ πάντως θεωρώ ότι η παρούσα Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να ταξιδέψει, να πάει στην Τουρκία φέτος για να συνομιλήσει με τους υπευθύνου στην Τουρκία για την κοινωνική, οικονομική κατάσταση στην χώρα και να καταστήσει σαφές ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Και αυτό να το καταστήσει και δημόσιο και να δείξει καθαρά η Επιτροπή μας ότι αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία δεν τα δεχόμαστε και μάλιστα να επιβραβευθούν κιόλα με μια ένταση της οικονομικής συνεργασίας. Αυτή τη θέση πρέπει να την καταστήσουμε σαφή και κατανοητή και στους πολίτες. Ενισχύοντα έτσι και τις δημοκρατικές εκείνε δυνάμει που ανθίσταται στην Τουρκία. Ταυτόχρονα όμως θεωρώ ότι για τη δική μας Επιτροπή είναι σημαντικό να καταστήσουμε σαφές ότι δεν μπορούμε να δρούμε και με τρόπο αντιφατικό. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλουμε κυρώσεις στην Ρωσική Ομοσπονδία μέσα σε, σε μια συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση. Ενώ δεν το κάνουμε αυτό απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να φανούμε και συνεπείς. Όταν λοιπόν επιβάλλουμε κυρώσεις, επίσης πρέπει να γνωρίζουμε και πώς θα βγούμε από αυτές. Νομίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή μας πρέπει να συζητήσει και ποια είναι η προοπτική. Αν δηλαδή τώρα προχωρήσουμε σε μια επικύρωση της οικονομικής συνεργασίας, πρέπει να γνωρίζουμε και πώς θα βγούμε. Αλλιώς δεν κάνουμε παρά μόνο πολιτική συμβόλων, η οποία δεν εξυπηρετεί ούτε εμάς ούτε τους ανθρώπους εκεί. Έχω άλλου δύο που ζητούν τον λόγο. Να είσαστε όμω σύντομοι, διότι αλλιώ ξεφεύγουμε από το χρονικό πλαίσιο. Κύριο κύριος Μπρούκνερ, ευχαριστώ. Προ δύο εβδομάδων πήγα στο ανατολικό μέρος της Τουρκίας, στο μέρος που κατοικούν οι Κούρδοι. Οι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είδα εκεί είναι απερίγραπτε. Δεν μπορώ να σα τι περιγράψω. Με λίγα λόγια μόνο. Υπάρχουν ολόκληρα τμήματα των πόλεων που κατοικούνται από, από Κούρδους και βομβαρδίστηκαν και κατεδαφίστηκαν. Πολλές εξοδικαστικές εκτελέσεις, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να δεχτούμε. Γνωρίζω άλλωστε από, την, από τον τουρκικό πληθυσμό ότι μέγα μέρος της στήριξης που έχει μεταξύ του τουρκικού πληθυσμού ο Ερντογάν οφείλεται και στην οικονομική ανάκαμψη. Εάν τώρα προχωρήσουμε σε νέα συμφωνία και πάμε να ενισχύσουμε στην οικονομική αυτή ανάκαμψη, ενισχύουμε άμεσα την στήριξη για τον Ερντογάν. Και νομίζω ότι όντω θα είναι ακριβώ το αντίστροφο μήνυμα αυτό, από αυτό που θέλουμε να δώσουμε. Κύριο Πάμπριξ, ευχαριστώ. Πολύ σύντομα αναφέρομαι σε προηγούμενα σχόλια. Κοιτάξτε, βεβαίω εφόσον μιλούμε για αναβάθμιση τη τελωνιακή ενώσεω, και των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, δεν μπορούμε να αποφύγουμε να εξετάσουμε και το συνολικότερο πλαίσιο. Αυτό είναι σαφές. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αποφύγουμε να πηδήξουμε σε άλλο ένα χαντάκι από μόνοι μας, συγκρίνοντας για παράδειγμα την Τουρκία με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, διότι εξακολουθεί να υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Μπορεί να μην μας αρέσει το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά να μην δυσμονούμε ότι επιβάλαμε διεθνείς εμπορικές και οικονομικές κυρώσεις στην Ρωσία, όχι επειδή φυλάκιζε τους αντιφρονούντες, αλλά λόγω της εξωτερικής επιθετικότητας απέναντι στην Ουκρανία, της κατάληψης και προσάρτησης της Κρυμαία. Νομίζω λοιπόν ότι η σύγκριση ανάμεσα στις δύο χώρες και στη στάση μας απέναντί τους για την ώρα, δεν, αυτή τη στιγμή δηλαδή, δεν είναι ορθή. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ο κύριος Πέτρος Σουμάλης, υπεύθυνο στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Yes, thank you very much. Uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρουσίαση και για τα έγγραφα εργασία τα οποία εκτιμούμε ιδιαίτερα. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ε, την, ε, να έχουμε μάλλον μια εκτεταμένη συζήτηση ε, μαζί του και με άλλους βουλευτές στην ομάδα παρακολούθησης. Οι εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία που χρονολογείται εδώ και 20 χρόνια ε, είναι ξεπερασμένη, πράγμα το οποίο μας κάνει να συζητάμε το θέμα της ανάγκης ανανέωσης των εμπορικών αυτών μας σχέσεων και έχουμε πει επανειλημμένα και επίσης αυτό το έχουμε δηλώσει και στην έκθεση προόδου για την Τουρκία που εγκρίθηκε από την Κομισιόν εχθές ότι έχουμε πει λοιπόν ότι η Κομισιόν εκπονεί την προπαρασκευαστική της εργασία για την πιθανή ε, παρουσίαση του σχεδίου διαπραγματευτικών οδηγιών για τα τέλη του τρέχοντος έτους. Όπως ξέρετε, η έκθεση προόδου ήδη παρουσιάστηκε χθε στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και θα συζητηθεί από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την επόμενη Δευτέρα. Ακούσαμε πολλά για τις τρέχουσε εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία, καθώς και για τα στοιχεία τα οποία λείπουν. Θα πρέπει οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση στην Τουρκία καταρχά να συγχρονίσει τη λειτουργία της υφιστάμενης Τελωνιακής Ένωσης και από την άλλη πλευρά να επεκτείνει το πεδίο της εμπορικής σχέσης σε νέους τομείς. Όταν λέμε για επέκταση του πεδίου εφαρμογή, σκεφτόμαστε διάφορους νέους τομείς για περαιτέρω βελτίωση και απελευθέρωση των συναλλαγών. Ε, σε τομείς όπως οι υπηρεσίες και οι κρατικές προμήθειες ε, που δεν καλύπτονται από την Τελωνιακή Ένωση, καθώς επίσης και φιλόδοξη προσέγγιση του γεωργικού τομέα. Αλλά όταν μιλάμε για επέκταση, Πρόεδρε, μιλάμε και για την επέκταση του ε, των κανόνων για το εμπόριο με Τουρκία ε, σε νέα σημεία γιατί δεν υπάρχουν ε, κανόνες για πολλά, πολλούς από τους τομείς αυτή τη στιγμή ε, και η επέκτασή τους και στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίες έγινε μεγάλος λόγος σήμερα. Βιώσιμη ανάπτυξη δεν υπάρχει στην Τελωνιακή Ένωση με την Τουρκία. Επίσης διατάξεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή για την αυξημένη διαφάνεια δεν υπάρχουν. Όλοι αυτοί οι κανόνες λοιπόν θα ήταν πολύ χρήσιμη προσθήκη στην ε, σχέση μας με την Τουρκία. Ξέρουμε πως σήμερα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και ότι υπάρχουν ε, πολλές περιπτώσεις όπου η συμμόρφωση της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της υπό Ένωση δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Ο εισηγητής αναφέρει και παραδείγματα και είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως υπάρχουν περισσότερες υποθέσεις από αυτές που αναφέρει ο εισηγητής, δηλαδή επιπλέον δασμοί επιβάλλονται και θα ήταν χρήσιμο πιστεύω για την έκθεση αυτή να δοθούν και άλλα παραδείγματα γιατί να μην πιστέψει κανείς πως πρόκειται για ένα μοναδικό παράδειγμα και βέβαια όταν ε, διαπραγματευόμαστε μια νέα εμπορική σχέση θα πρέπει να επιμείνουμε για αυτά ε, τα ε, ήδη υπάρχοντα προβλήματα όπως αυτή οι εμπορικοί περιορισμοί. Ανέφερα λοιπόν πως η Κομισιόν συνεχίζει την προπαρασκευαστική της εργασία ώστε να μπορεί να υποβάλλει τη θέση της στο τέλος του έτους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανερχόμαστε στον εισηγητή μας. Παρακαλώ. Και ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για τις ε, τοποθετήσεις σας. Παραλαμβάνω τη βούλησή μου. Είναι να ξεκινήσουμε μαζί όλοι μια συζήτηση που θα καταλήξει σε ένα όσο το δυνατόν πιο συνενετικό έγγραφο, γιατί είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και βεβαίως δεν θέλει κανείς να συνεχίσει το business as usual. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Στις επόμενες ημέρες λοιπόν θα επικοινωνήσω και με τα γραφεία σας έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ε, επεξεργασία του εγγράφου για τις προσεχείς μας συναντήσεις. Έχουμε 28-29 Νοεμβρίου τη συνεδρίαση στην οποία θα εστιαστούμε ιδιαίτερο στην ανταλλαγή απόψεων με εμπλεκόμενους ε, παράγοντες τόσο Ευρωπαίους όσο και Τούρκους. Είναι πολύ σημαντική εν ώψη της επίσκεψής μας στην Τουρκία και βεβαίως σας καλώ όλους να είστε παρόντες σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτή τη συνεδρία. Σας ευχαριστώ. Herzlichen Dank. Σας ευχαριστώ. Άρα κλείνει και το σημείο 14. Και τώρα πάμε στις ψηφοφορίες. Που βέβαια οι συνάδελφοι υπολογίζουν πως θα ξεκινήσουν στις 10, άρα διακόπτω μέχρι τις 10 η ώρα ακριβώς, αλλά 10 ακριβώς.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen Sie bitte Platz. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τώρα και σας παρακαλώ να καθίσετε στις θέσεις σας. Good. Wir haben gestern ja die Änderung der Tagesordnung beschlossen. Λοιπόν, χθε αποφασίσαμε την αλλαγή τη ημερήσια διάταξη κατά στο ώστε το σημείο 15 να ε, ψηφιστεί μετά το 21, δηλαδή θα έρχεται τελευταίο στον κατάλογο των ψηφοφοριών μα και ψηφίζουμε πρώτα το 16 σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχέση και συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας μεταξύ ευρωπαϊκή ενωση και Ουσβεκιστάν. Πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, ας κάνουμε ένα δοκιμαστικό παρακαλώ για να δούμε ότι λειτουργούν όλα τα μηχανήματα. Έχετε τις κάρτες σας ελπίζω να λειτουργούν και όλα. Αρχίζει τώρα η δοκιμαστική ψηφοφορία.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 Ωραία, λοιπόν, προχωρώ στην ψηφοφορία για τη σχέση με το Ουσμπεκιστάν. Συμβαστική τροπολογία 4, παρακαλώ. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 22, υπέρ, κατά. Αποχές, απερίφθη. Συμβαστική 6, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 28 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορεί να έχει εγκριθεί, ας επαληθεύσουμε την 27. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ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 απερίφθη 15 υπέρ κατά αποχές ε, απερίφθη 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπάρχει μόνο ένα υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την ένα αρχής ψηφοφορία Πέρας. Και εγκρίνεται. Δύο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1 από την άφετη τώρα χρωματότηση. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέμπτη παράγραφος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έβδομη παράγραφος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ενάτη παράγραφος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα. Ενδεκάτη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δωδεκάτη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκάτη τρίτη παράγραφος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά Δεκαπέντε, γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε μια γραμμή, δεν την είχαμε ψηφίσει, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα. Ηλεκτρονικά. Πέρασε της ψηφοφορίας. Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίνεται και συγχαρητήρια και ευχαριστία στην εισηγήτρια. Τώρα, σημείο 17. Ουσιαστικά είναι το ψήφισμα που ακολουθεί το προηγούμενη ψηφοφορία. Ε, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και πάλι εγκρίνεται με πολύ. Ισχυρή πλειοψηφία, συγχαρητήρια. Και πάω στο σημείο 18. Συνένεση, σύμφωνη γνώμη μάλλον για την ε, εταιρική οικονομική σχέση με την Κάνα, ηλεκτρονική ψηφοφορία, μοναδική και την ε, και κυρίσω την έναρξή τη. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια. Σημείο 19 τώρα, ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβαστική 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται πέρας άλλη μια ισχυρή πλειοψηφία εγκρίνεται και συγχαρητήρια και πάμε στο σημείο 20 ετήσια έκθεση χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ τη 13 13 λοιπόν παραλαμβάνουμε υπέρ Κατά. Αποχές. Και επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές Α κάνουμε μια επαλήθευση. Όπως είπα, τροπολογία 16. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τελική δε ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά αρχίζει Πέρας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Δεν μπορώ να δώσω προσωπικά στον εισηγητή τα συγχαρητήρια διότι νομίζω ταξιδεύει στη Γαλλία. Ερχόμαστε στο 21. Με, πριν από την ψηφοφορία έχουμε μια πρόταση για προφορική ερώτηση. Όπω άλλωστε συμφωνήσαμε χθε με του συντονιστέ. Θα την ψηφίσουμε. Ψήφι υπέρ της προτάσεω προφορικής ερωτήσεω. Παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Και ακολουθεί η έκθεση. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές Ας επαληθεύσουμε καλύτερα. Τροπολογία 12. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία, μάλλον συγγνώμη, τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές. Το Λαϊκό Κόμμα για την τροπολογία 24 είστε κατά. Ας επαναλάβουμε την ψηφοφορία για να είμαστε πιο σίγουροι. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε 25 αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας απερίφθη τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβατική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία που γίνεται ηλεκτρονικά αρχίζει. Πέρασε. Με μεγάλη πλειοψηφία, όπως βλέπετε. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Έρχομαι στο 15 τώρα. Την μακροοικονομική υποστήριξη προς την Ιορδανία. Όπως γνωρίζετε, επιτύχαμε συμφωνία με το Συμβούλιο Υπουργών σε εντατικό τριμερή διάλογο και το αποτέλεσμα το έχετε μπροστά σας για ψήφιση και αρχίζει η σχετική ψηφοφορία. Πέρας. Mm. Με μεγάλη λοιπόν πλειοψηφία εγκρίνεται. Άρα μπορεί να απελευθερωθεί, να το κονδύλια δηλαδή για την μακροοικονομική στήριξη. Έρχομαι τώρα στο υπαριθμό 22. Έκθεση για τις ομάδες παρακολούθησης, monitoring δηλαδή, που έχουν ήδη διεξαχθεί. στις 12 Οκτωβρίου διεξήχθη monitoring group για την συμφωνία TTIP για το 15ο γύρο και, και ορισμένες συνομιλίες stock taking δηλαδή διαπίστωση της προόδου μέχρι τώρα ενημερωθήκαμε πάντοτε με όλες τις σχετικές δυσχέρειες Και τώρα βέβαια ακόμα περισσότερο, περισσότερες δυσκολίες αναμένονται με την αλλαγή κυβερνήσεως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έγινε στις 13 Δεκάτου άλλη monitoring group για τον 20ο γύρο. Για τη δεύτερη τροποποιημένη προσφορά από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητής όμως είναι απόν. Έγινε και ένα monitoring group για την Ανατολικοαφρικανική κοινότητα στις 17 δεκάτου αυτό. Ο κ. Σόλτς όμως είναι παρόν και ίσως θέλει να πει κάτι σχετικά. Helmut Monitoring Group East African Community. Έγινε ανταλλαγή απόψεων με τους πρέσβεις της Ανατολικοαφρικανικής κοινότητος. Ο πρέσβης της Τανζανίας μας ενημέρωσε ότι μέχρι την επόμενη διάσκεψη των Προέδρων δεν υπάρχει σαφήνεια σε ό,τι αφορά τις θέσεις των πέντε χωρών για τη διαδικασία και μάλλον θα χρειαστεί να περιμένουμε λοιπόν να διεξαχθεί αυτή η διάσκεψη τον Δεκέμβριο και μετά η ενημέρωση θα γίνει τον Ιανουάριο. Για την ώρα λοιπόν δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με το ποιες θα είναι οι τελικές θέσεις των χώρων αυτών σχετικά με την συνέχιση και ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Α, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, έτσι είναι. Στις 17 Οκτωβρίου, Ουκρανία, Monitoring Group. Ο κύριος Βαλένσα είναι ε, διαρκής συγητής. Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε Βαλένσα. Συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό, που είναι πρόθυμος να προχωρήσει με τα ATM. Θα χρειαστεί να εξετάσουμε βέβαια την εφαρμογή της συμφωνίας από την αρχή του χρόνου. Ήδη γίνονται υπολογισμοί των επιπτώσεων. Είναι προφανές όμως ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αναλύσουμε την κατάσταση, για να γνωρίζουμε τι στάση ακριβώς θα τηρήσουμε. Προτείνω λοιπόν για τη συγκεκριμένη υπόθεση να προχωρήσουμε αργά, να είμαστε δηλαδή βέβαιοι ότι αναλύουμε όλα τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα των προτάσεων που έχουν ήδη κατατεθεί. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Λάγκερ. Monitoring Group τώρα για την Mercosur. Ο κύριος Σάλβα ε, φαίνεται πως είναι απόν. Επρόκειτο για ανταλλαγή σχετικά με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις. Γνωρίζουμε ότι μετά από ένα μακρό, μια μακρά παύση στις διαπραγματεύσεις με την Mercosur τώρα ε, έρχεται μια επιτάχυνση και το πρόσημα είναι θετικό. Στις 19 Δεκάτου διεξήχθη Monitoring Group για την Κεντρική Ασία. Ιδίως δε για θέματα του Ουσμπεκιστάν. Μόλις τα εγκρίναμε. και καταστήσαμε σαφή έτσι την θέση του Κοινοβουλίου. Στις 20 Οκτωβρίου, Monitoring Group για την Ιαπωνία. Γνωρίζετε ότι μετά από τις εκλογές για την Άνω Βουλή στην Ιαπωνία, οι διαπραγματεύσεις έχουν λάβει νέα όθηση και οι προοπτικές είναι καλές για τελική σύναψη συμφωνία με την Ιαπωνία. Είναι θετική η κατεύθυνση. Εάν δηλαδή δεν υπάρξει πρόοδος στην ε, συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, η Ιαπωνία θα είναι μάλλον διατεθειμένη να έρθει σε κάποια συμφωνία με την Ευρώπη. Monitoring Group επίσης για το Μεξικό. Όμως είναι εδώ ο συγκεκριτής, ο κ. Μωυσά. Ευχαριστώ. Όντω ε, σκέφτηκε η ομάδα παρακολούθηση πριν δύο μέρε Έχουμε και ένα δεύτερο γύρο που θα γίνει στο, το Νοέμβριο στο Μεξικό. Ο πρώτος γύρος, όπως θα αναμένα, ήταν πιο τυπικός. Προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Ε, πάντως, ε, προετοιμάζοντας τον δεύτερο γύρο, η Κομισιόν έχει ήδη προετοιμάσει και έχει έρθει σε επαφή με τα κρατημέλη για προτάσεις για εννέα τομείς ε, κανόνες προέλευσης, δημόσιες προμήθειες, προτεσίλες και διάφορα και διάφορα άλλα. Θα είναι δηλαδή ουσιαστικός αυτός ο γύρος. Οι Μεξικανοί έχουν ήδη δεσμευθεί να στείλουν κάποιες γραπτές προτάσεις και για τους ε, φόρους. 22 μέχρι 25 Νοεμβρίου θα μιλήσουμε για τους δύο Τομεί από τις 20 για που εμπίπτουν στη διαπραγμάτευση και βέβαια αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να διαλύσει την ναύτα τότε τα κίνητρα για τους Μεξικανούς σε αυτή τη διαπραγμάτευση θα αλλάξουν τελείως. Και θα πρέπει και εμείς να αξιολογήσουμε τις δικές μας φιλοδοξίες και προτεραιότητες σε αυτό το νέο κόσμο που προκύπτει, που αναδύεται. Για την ώρα έχουμε σχετικά αργούς ρυθμούς διαπραγματεύσεων. Έχουμε και κάποια εργασία ανάμεσα στις ε, ε, συνόδους. Πολλά θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει σε αυτό το δεύτερο γύρο όσον αφορά τη φιλοδοξία και την ταχύτητα με την οποία θα δουλέψουμε και οι δύο πλευρές. Γιατί και εκείνοι θα χωνεύουν σιγά σιγά τις τα αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και έτσι ακούσαμε τα περισσότερα τουλάχιστον πεπραγμένων των ομάδων παρακολούθησης των monitoring groups. Υπενθυμίζω συναδέλφους ότι είναι κομμάτι σημαντικό της δουλειά μας και έτσι είναι καλό να έχουμε την ευκαιρία της ανταλλαγής απόψεων στους τομείς που μας ενδιαφέρουν γιατί ευκολύνει και τη δουλειά μας. Μπορούμε έτσι να την κάνουμε και πιο σοβαρά. Και έτσι φτάνω στο σημείο 23, αγαπητοί συνάδελφοι. Το σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σημερινή συνεδρίασης. Ε, τα συμπεράσματα σχετικά με την Συμφωνία Εμπορικών Σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. ΣΕΤΑ. Και είχαμε υπολογίσει για σήμερα μια συζήτηση μεταξύ συναδέλφων Επιτροπής και Συμβουλίου. Ως προς τον, τους δύο τελευταίους έχουμε το εξής πρόβλημα. Ότι έχει κλείσει το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι δεν μπορούν να έρθουν οι δύο υπεύθυνοι, ο Διευθυντής και επικεφαλής διαπραγματευτής, διότι είναι αποκλεισμένη από τους, ε, τους εργάτες χαλιβουργίας που διαμαρτύρονται. Έτσι, από την Επιτροπή δεν μπορούμε να δούμε κανέναν και για το Συμβούλιο και την Προεδρία. Πάλι δεν μπορούμε να έχουμε κανέναν γιατί είναι απασχολημένοι στην προετοιμασία του Συμβουλίου. Πάντω εκπροσώπηση τη Προεδρία έχουμε, απλώ δεν έχουμε κορεπέρ. Και ελπίζω να μπορέσουμε να ακούσουμε, να δούμε μάλλον σύντομα και τους εκπροσώπους τη Επιτροπής. Η συμφωνία όπως γνωρίζετε. Υπεγράφει στις 30 Οκτωβρίου, Κυριακή. Με μια κάποια καθυστέρηση σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Αλλά από 30 Οκτωβρίου, 30 Οκτωβρίου έχουμε αυτή τη συμφωνία. Ένα μέσον. Ένα νομοθέτημα που έχει υπογραφεί από την κυβέρνηση του Καναδά, τα 28 κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που συνοδεύεται από 28 γραπτές δηλώσεις. Ένα πακέτο το οποίο έχει διαβαστεί εντωμεταξύ στο Κοινοβούλιο και με βάση αυτό ξεκινούμε την επίσημη διαβούλευση. οι συνομιλίες για τις συνοδευτικές του κειμένου δηλώσεις είναι καταρχάς το μέσο και ιδιαίτερα εδώ για τους συναδέλφους του Κοινοβουλίου ε, η πρόταση την οποία υποστήριξαν, η λύση την οποία υποστήριξαν έτσι ώστε να διευκρινιστούν διάφορα σημεία τα οποία θεωρήθηκαν χρήσιμα για την περαιτέρω συνεργασία των εταίρων και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν χρήσιμο θα ήταν χρήσιμο να γίνει να δοθούν οι διευκρινήσεις στα θέματα αυτά. Ως πρόεδρος Επιτροπής Εμπορίου πάντως δεν είμαι σε θέση να δεχθώ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να μένει εκτός της ε, διαπραγματεύσης του Κοινοβούλου να μην έχει κατάλληλη ενημέρωση δηλαδή. Μας απέκλεισε το Συμβούλιο, ενώ θα έπρεπε να μας ενημερώνει τακτικά για τα διάφορα στάδια της διαπραγμάτευσης. Το έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα αυτό, ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται για κάθε στάδιο της διαπραγμάτευσης. Αυτά. Ως προς τι επικρίσει από πλευράς μας, δεν είχαμε αυτή την ενημέρωση. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια σε συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή να βελτιώσουμε τη διάσταση αυτή. Τώρα έχουμε ένα νομοθέτημα, μια συμφωνία, μια δήλωση με τις δηλώσεις της που αποτελούν ένα σύνολο και που θα μας παρουσιάσει τώρα ο εισηγητής μας κύριος Πάμπριξ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Βεβαίω λυπούμε που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τον διαπραγματευτή μας Πετριτσιώνη εδώ, γιατί πολλές ερωτήσεις, ε, πολλά θέματα πρέπει να αποσαφηνίσουμε με τον, την Επιτροπή και με εκείνον τον ίδιο, γιατί είναι ένας από τους πιο έμπειρους διαπραγματευτές σε αυτήν ε, την υπόθεση. Εν γέννη, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι που επιτέλους υπογράφηκε αυτή η συμφωνία με τον Πρωθυπουργό Τρουντό, αν και δεν ήταν ε, στρωτός ο δρόμος ε, προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Θα πρέπει να μείνουμε λοιπόν, να επιμείνουμε στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, σε αυτά που έχουμε ήδη δηλώσει, ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα με, την ταχύτητα, ε, με ταχύτητα στην συζήτηση εδώ για τα μέρη που έχουν απομείνει για αυτή τη συμφωνία, καθώς και να προχωρήσουμε ε, στην επικύρωση από πλευρά του Κοινοβουλίου μας, διότι για πολλού, πολλά κομμάτια αυτής της ε, συμφωνίας είχαμε αρκετές πληροφορίες, ωστόσο, όπως μάλλον θα θα θέλουν να θέσουν ερωτήσεις οι συνάδελφοι στον κύριο Πετριτσόνε για το πώς γενικά έγιναν οι ε, ad hoc συνεδριάσεις με το Βέλγιο και ένα κομμάτι του Βελγίου πώς διοργανώθηκαν και τα λοιπά. Νομίζω πως <laughs> πρόκειται για μια λίγο αμφισβητήσιμη διαδικασία και θα θέλω να ρωτήσουν τον κύριο Πετριτσόνη πώς γίνανε όλα αυτά. Επίσης έχουμε μεταβεί σε ένα νέο είδος δηλώσεων διότι δεν είναι 100% σαφές το πού θα τοποθετήσουμε και πώς τις βλέπουμε μέσα σε όλη αυτή τη γενική συζήτηση και δίκτυο συζήτησης εντός του Κοινοβουλίου. Νομίζω λοιπόν πως αυτές οι ερωτήσεις ήθελα να θέσω στον κύριο Πετριτσόνη όταν θα φτάσει Πάντως η γενική γραμμή μου και η γραμμή του κόμματός μου παραμένει απαράλλακτη. Πρέπει να προχωρήσουμε όσο γίνεται ταχύτερα, ιδιαίτερα θα πρέπει αυτό να γίνει λαμβάνοντας υπόψη την γενική κατάσταση προόδου των υποθέσεων αυτών στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ιφίλιο θα πρέπει η υπογραφή ε, αυτή τη συμφωνία να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να σφραγιστεί μάλλον όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μόλι μου είπαν ότι έχει ξανανοίξει το κτίριο, έχει απεμπλακεί και ότι ο Μαουρίτσιο έρχεται. Ο κύριος Μόησα, εν τω μεταξύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ελπίζω πως ο Μάουρο θα έρθει σύντομα Ελπίζω πως θα μπορέσει να μας απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να πω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα από τη δική μου πλευρά και πιστεύω και οι περισσότεροι από τους συναδέλφους τα βλέπουν παρομοίως. Πολλές αμφιβολίες και άγχος επικράτησαν αυτή την, για αυτή την συνθήκη. Δεν οφείλονταν στον λαϊκισμό ή σε παράξενη μυστική ατζέντα, όπως είπαν κάποιοι, μάλλον πήγαν να πούν κάποιοι, να προτείνουν κάποιοι. Απορρίπτω ε, την ιδέα ότι οι συνάδελφοί μου είναι λαϊκιστές. Είναι φυσιολογικό να έχει κανείς ερωτήσεις και αμφιβολίες και να προσπαθεί να τις αποσαφηνίσει. Δυστυχώς η διαφάνεια δόθηκε για πολλά από αυτά τα θέματα, έχουμε όμως κάποια ακόμα και θα έρθω σε αυτά σε λίγο, αλλά αυτή η σαφήνεια δυστυχώ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό εκτός αυτού εδώ του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι οδυνηρό, αλλά είναι και κομμάτι της ευρύτερη δημοκρατικής διαδικασίας που έχουμε στην Ευρώπη, δηλαδή Περισσότερη συζήτηση θα πρέπει να έχει γίνει εδώ για αυτή τη συνθήκη με τους συναδέλφους, ώστε να απαντήσουμε και στις ερωτήσεις και στις αμφιβολίες. Τώρα, είμαστε σε αυτή την κατάσταση, έχουμε ένα μακρύ κατάλογο δηλώσεων παρατήμα της συνθήκης και πρέπει να υπάρξει σαφήνεια για την ε, καθεστώς αυτών των δηλώσεων πώς αυτές σχετίζονται με τη ΣΥΤΑ. Θα είναι ενδιαφέρον και ελπίζω ότι θα ακούσουμε από τον Μάωρο τι σκοπούς έχουν, τι πώς σχεδιάζουν να ε, αντιμετωπίσουν και να θέσουν σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα που περιλαμβάνεται. Πρόγραμμα εργασίας στην ουσία είναι. Γιατί πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα αντιμετωπίσει η Κομισιόν αυτό το θέμα Επίσης θα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα δουλέψει η ρήτρα ασφαλείας για τη γεωργία στην οποία αναφέρεται το Βέλγιο που θα μπορούσε εκεί να υπάρξει κάποια ένταση εκεί ανάλογα με την θέση του, του Βελγίου ή αν αυτό θα εμποδίσει τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έπειτα, συνάδελφοι, δεν θέλω να τώρα δω να πω όλε τι ερωτήσει που θέλετε να, βάλετε, να θέσετε κι εσεί. Το... Είμαι σίγουρο ότι θα τι θέσετε στο Μαουρό όταν θα φτάσει. Πάντω υπάρχει ένα σημαντικό σημείο. Και στο, στα όσα λέει που Μπορεί να έχουμε αρνητικές πτυχές στο εμπόριο, πώς θα καταπολεμήσουμε ακόμα ή πώς θα σχηματίσουμε, την, ε, πώς θα επηρεάσουμε την ε, παγκοσμιοποίηση, ε, πώς θα την ακυρώσουμε, όπως λέει ο Τραμπ, και το, πώς θα ακυρώσει την ΑΦΤΑ, λέει. Εν πάση περιπτώσει, είναι σωρό άλλα αρνητικά πράγματα. Πάντως είναι σημαντικό για τους συναδέλφους και για τους Καναδούς εταίρους μας να έχουμε σαφήνεια για τη θέση της ΣΥΤΑ και τον τρόπο εφαρμογή τη εφαρμογής της όσο γίνεται νωρίτερα. Να το, να το αποφασίσουμε σε αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα ως μια αξιοπρεπή αντίδραση στα, στα όσα συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο και στι αμερικανικέ εκλογές. Μπορεί να συμφωνούμε ή όχι με ορισμένα πράγματα στην συνθήκη. Πάντως πρέπει να δώσουμε τη γνώμη μας για την ΣΕΤΑ. Αυτό είναι καθήκον μας. Είναι θέμα αξιοπρέπειας απέναντι στους Καναδούς εταίρους, οι οποίοι πιθανόν είναι να, απομονωθούν αρκετά στη Βόρεια Αμερική, αν ο Τραμπ παίρνει τον εαυτό του σοβαρά και θελήσει να κάνει έστω και τα μισά από αυτά που είπε ότι θα κάνει, ο Καναδάς μάλλον θα θελήσει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια γενιά. θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Λοιπόν, νομίζω πως ε, θα πρέπει αυτό να το σκεφτούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση προς χάνη της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, άσχετα με το τι θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. ECR Κάμπελο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συνεχίσω για τα όσα είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Όντως το ότι εξελέγει ο Τράμπα θα αλλάξει την κατάσταση για το ελεύθερο εμπόριο αρνητικά και όλη η ατμόσφαιρα, το νέο κλίμα για το ελεύθερο εμπόριο θα αλλάξει. Το TTIP ε, ε, είναι σε κίνδυνο. Έχει μιλήσει ήδη για την ΑΦΤΑ και αυτό θα έχει επιπτώσεις και για τον Καναδά αν ο πρόεδρος Τραμπ όντως φύγει από την ναύτα. Έχει λοιπόν επιπτώσεις και για την ΣΕΤΑ. Είναι πολύ καλή συμφωνία, είναι η καλύτερη που έχει ποτέ κάνει η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλές αυτό που ίσως να έχει χαθεί στο κείμενο είναι ότι είναι η, σοβαρό... η μεγαλύτερη συμφωνία που έχουμε ποτέ κάνει με έναν μεγάλο εμπορικό μας εταίρο. Πράγμα που έχει μεγάλη σημασία το ίδιο. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε γιατί τελείως θα καταντήσουμε περίγελος. Ήδη γίναμε περίγελος λόγω της ε, αντίδρασης της Βαλωνίας. Εντάξει, είναι θέμα δημοκρατίας, οκ, okay, αλλά σχεδόν χάθηκε η συμφωνία και βρεθήκαμε σε πολύ δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να προχωρήσουμε και να δούμε ποια είναι τα ωφέλη. Πρέπει όντω να το ψηφίσουμε το Δεκέμβριο, προσωρινώς να εφαρμόσουμε την συμφωνία από τις αρχές του επόμενου έτους και να συνεχίσουμε. Ε, και να δώσουμε το καλό παράδειγμα στον κόσμο. Ευχαριστώ εκ μέρους των ε, φιλελευθέρων κυρία Σχάκη. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Δεν παρακολουθώ πια καν τις ευκαιρίες που είχαμε να συζητήσουμε τη ΣΕΤΑ. Κάθε ευκαιρία φυσικά είναι ευπρόσδεκτη. Κάθε ευκαιρία να συζητήσουμε τη ΣΕΤΑ και τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα αναλάβουμε τις σχετικές ευθύνες για την υλοποίησή της. Έχουμε θίξει μια σειρά από ζητήματα που με χαρά βλέπω ότι καταγράφονται στο τελικό αποτέλεσμα. Συμφωνώ, όπως είπε ο κ. Μόησα, ότι δεν μπορούμε να σοπίσουμε όταν βλέπουμε ζητήματα στα οποία πρέπει να ε, αντιδρούμε. Από την άλλη πρέπει να δούμε και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες. Όταν έχουμε έναν αποτρόπαιο πόλεμο ε, να μένεται στη Συρία ή τις εξαγωγές όπλων προς αυτούς παραβιάζουν κατά τον χειρότερο δυνατό τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν βλέπω να κατεβαίνει κανείς στον δρόμο για να τους υπερασπιστεί, για να υπερασπιστεί αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά για τον Καναδά κατεβαίνουν στον δρόμο και δεν το καταλαβαίνουν. Ένα τελευταίο λοιπόν κομμάτι της πορείας για τις διαπραγματεύσεις ε, αυτές αποδείχθηκε αρκετά ε, δύσκολο, αρκετά δύσβατο πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα για να μην ε, το ξεβατιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να ετοιμάσουμε κατά τρόπο πιο σωστό, πιο καλό, πιο επαγγελματικό προσεχή συμφωνίες. Είναι καλή η συμφωνία ΣΕΤΑ για όλους ε, και πρέπει το ταχύτερο δυνατό να αντλήσουν τα ωφέλη της από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και πιστεύω ότι και εμείς πρέπει πρόεδρε να καταγράψουμε αυτά τα οποία είδαμε να συμβαίνουν κρίσιμες συζητήσεις ε, αναπτύχθηκαν με απόλυτο αποκλεισμό της ε, Επιτροπής μας. Είδαμε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να λαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες για τις οποίες είμαστε σε πλήρη άγνοια. Δεν ξέρω αν είχε μαζί με εσάς κάποιες διαβουλεύσεις, αλλά ξαφνικά τον είδαμε να αναδεικνύεται σε ρόλο, να, να αναλαμβάνει ρόλο και ε, αρμοδιότητες δικές μας κανονικά σε αυτές τις διαδικασίες. χρειαζόμαστε επίσης σαφείς εντολές σε σχέση με τη δράση των κρατών μελών το ρόλο των διαφορών θεσμικών οργάνων και ιδιαίτερα πρέπει να υπογραμμιστεί η υποχρέωση τήρησης των συνθήκων. Επίσης θέλουμε σαφείς κανόνες για το ποιος μπορεί να αναλάβει μέτρα μετριασμού των συνεπειών ε, ενδεχομένων αρνητικών συνεπειών συγκεκριμένα του εμπορίου. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω έπρεπε να έχει συζητηθεί και η χθεσινή συζήτηση που έγινε για το διεθνές εμπόριο και αν κάποιοι συνάδελφοι δεν ήταν παρόντες σου ενημερώνω, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και οι διάφορες ομιλίες που ακούσαμε πολύ ε, ενημερωτικές. Πάντως αυτό που ιδιαίτερα ακούστηκε ήταν ότι θα πρέπει να γίνεται πιο ξεκάθαρα η συζήτηση για το τι μπορούν να επιτύχουν και ε, τι δεν μπορούν να επιτύχουν οι εμπορικέ συμφωνίε, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του φόβου έχει να κάνει με την άγνοια τη πραγματικότητα και σε αυτό έχουμε εμεί ρόλο να διαδραματίσουμε, να εξηγούμε τι είναι δυνατόν και τι δεν είναι. Ιδάλω θα μπλέκουμε όλο και σε χειρότερα προβλήματα. Και επίσης ε, πολύ περισσότερο τώρα από τη χτες ή από πέρσι είναι απαραίτητο να υπογραμμίσουμε πόσο σοβαρή δύναμη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματευτής πόσο ισχυρό ρόλο έχει και στο παγκόσμιο σκηνικό και με ένα νέο εκλεγέντα πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος έχει τουλάχιστον ε, της λόγης ε, επιδείξει την ε, άγνοιά του, πάση περιπτώσει το ότι παραγνωρίζει τη σημασία των διεθνών σχέσεων. Έχει έρθει η ώρα για μας να αναλάβουμε πιο ισχυρό ρόλο με σαφείς προδιαγραφές, με κανόνες, με πρότυπα με εξυγχρονισμό των συμφωνιών που είχαμε μέχρι τώρα και πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε σοβαρές απαντήσεις σε αυτούς που θεωρούν ότι το εμπόριο μπορεί να είναι ένας τρόπος να καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να αποδιαρθρωθούν οι αξίες που χαρακτηρίζουν τις συμφωνίες που έχουμε οικοδομήσει ουσιαστικά από το τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε σαφεί και απέναντι σε αυτού που εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι μπορούμε να συνεχίζουμε επαόριστον τι διαπραγματεύσει χωρί καλή μια κατάληξη. Μια διαδικασία ολοκληρώνεται. Χαίρομαι που ολοκληρώθηκε και δεν πρέπει να λησμονούμε τι διακυβεύεται και τι ουσιαστικά μα απασχολεί όλου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σάκε, ο Μάουρο Πετιτσίνο ήρθε, έφτασε μπόρεσε και πέρασε μέσα από το φράγμα των χαλιβουργών. Έχουν θέσει ερωτήσεις οι προηγούμενοι ομιλητές, ιδίως όσον αφορά την διαδικασία αναζήτησης των περιγραφών του καθεστώτος που έχει το έγγραφο, καθώς και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα των περαιτέρω εργασιών, ιδίως για το σύστημα ICS, και τι σημαίνουν οι ρήτρε διαφύλαξης για την γεωργία από τη βελγική πλευρά γενικότερα. Αυτές είναι βασικά οι ερωτήσεις που τέθηκαν ως τώρα, αλλά σίγουρα θα έλθουν και άλλες. Αν Μαρή Μινέρ από την ε, Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε εδώ ε, θα ήθελα πρώτα να διαμαρτυρηθώ για το γεγονός ότι η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου δεν κάνει τη δουλειά της και δεν ψηφίζει, δεν προτείνει ψήφισμα. Η ΣΕΤΑ δεν είναι μια απλή συμφωνία. Έχει βαθύτατες επιπτώσεις στα δικαιικά μας συστήματα στη δημοκρατία μας, στα τρόφιμα που καταναλώνουμε και ούτω καθεξής. Εκτός από αυτό, το γερμανικό ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο επισημαίνει σε απόφασή του ότι θα υπάρχουν βαρύτες επιπτώσεις από την εφαρμογή της συμφωνίας. Και από πλευράς καναδικής υπάρχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με την συμφωνία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να απασχολήσουν τους βουλευτές και να τοποθετηθούν. Υπάρχουν και πολλά νομικά θέματα τα οποία δεν έχουμε εξετάσει καθόλου. Για παράδειγμα, εάν το σύνολο της συμφωνίας είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό δικαιικό σύστημα και η προσωρινή ισχύ του κλπ. Προσωρινή ισχύ της συμφωνίας θα χρειαστεί να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για τη συμφωνία με την Σιγκαπούρη και βεβαίω πρέπει να πούν τη γνώμη τους και οι ευρωβουλευτές. Και εν τέλει τίθεται και το θέμα ε, κόστους οφέλους. Υπάρχουν μελέτες και υπάρχουν και από την Αυστριακή Ένωση Εργαζομένων πολλές επιφυλάξεις και πολύ σοβαρά ερωτήματα που ξεπηδούν σχετικά με την απασχόληση και υπάρχουν και νέες πολιτικές εξελίξεις. Και πολλοί του έχουν ταχθεί κατά των ε, εμπορικών συμφωνιών. Σας θυμίζω και τις σημαντικές επιπτώσεις του Brexit. Η Μεγάλη Βρετανία είναι και με απόσταση μεγάλη ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Καναδά. Επαναλαμβάνω ότι οι ευρωβουλευτές πρέπει να τοποθετηθούν για όλα αυτά. Και παρόλα αυτά, οι περισσότερες πολιτικές ομάδες δεν θέλουν να επιτρέψουν να ε, καταθεί πρόταση ψηφίσματος από την Επιτροπή μας. Για ποιο λόγο, γιατί φοβούνται τόσο πολύ να αλλάξουν έστω και ένα γράμμα της Συμφωνίας ΕΤΑ, παρόλο που αυτό θα βοηθούσε να βελτιωθεί, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε είπε το εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι κοινοβούλιο, είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να φέρει το όνομα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι βεβαίω κοινοβούλιο όπω το δικό μα, το Ολλανδικό Κοινοβούλιο δηλαδή. Ούτε και η Κομισιόν δεν είναι κυβέρνηση. Και όπω η Κομισιόν δεν είναι κυβέρνηση, έτσι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι όπω τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχει τελείω διαφορετικέ αρμοδιότητες. Αυτά λέει ο, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός, τα είπε μάλιστα την 1η Νοεμβρίου στην Ολλανδική Γερουσία. Στο μεταξύ εγώ έχω ακούσει ότι η εμπορική πολιτική γίνεται σταθερό θέμα στην ημερήσια διάταξη και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Αυτό δείχνει ότι δεν εμπιστεύονται πλέον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν αρκεί λοιπόν να εξετάσουμε επιφανειακά την Συμφωνία ΣΕΤΑ. Χρειαζόμαστε ένα πλήρες ψήφισμα. Αυτό μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αλλά γιατί άραγε να επιταχύνουμε τώρα όταν οι διαπραγματεύσεις έχουν πάρει τόσα χρόνια. Η κριτική που ασκείται είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει δημοκρατική διαδικασία. Εδώ, ε, κοιτάξτε, έχω να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα και προς το κοινό. Πρώτα-πρώτα, εδώ είμαστε δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα και έχουμε καθαρά την αρμοδιότητα για το εμπόριο. Και εκπληρούμε τα καθήκοντά μας με πολύ καθαρό τρόπο, αναλύουμε κάθε εμπορική συμφωνία με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο. Ορισμένες φορές δεχόμαστε τι εμπορικέ συμφωνίε, ορισμένε άλλε φορέ, όπω πράξαμε και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο τι απορρίπτουμε. Αυτή είναι η δική μα ευθύνη και εμεί ω δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα, θεσμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπληρώνουμε τα καθήκοντά μα. Με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιδημοκρατικό το ό,τι συμβαίνει εδώ. Δεύτερο, οι πολιτικέ ομάδε, οι κοινοβουλευτικέ ομάδε, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισαν να μην κατατεθεί ψήφισμα από την Επιτροπή μας, αλλά από τις πολιτικές ομάδες στην Ολομέλεια, ώστε να αναμειχθούν όλοι οι ευρωβουλευτές. Ούτε αυτό το βρίσκω αντιδημοκρατικό. Πρόκειται για δημοκρατική διαδικασία, εφόσον μάλιστα επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των ευρωβουλευτών, όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων, ώστε θα ε, κατατεθεί ψήφισμα, θα ψηφιστεί ψήφισμα και επομένω θα υπάρχει θέση του ε, δημοκρατικά εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά λοιπόν για να καταστεί σαφές περί τίνος πρόκειται. Ας ακολουθήσει τώρα η κυρία Μπιγκίν. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ο Γιάννη Ξαντό δεν είναι παρόν, αλλά τον εκπροσωπεί η Κέλλερ. Ευχαριστώ. Όντω η πλειοψηφία αποφάσισε να μην καταθέσει ψήφισμα. Αλλά έχουμε αυτό το joint instrument, όπως επίσης και τις δηλώσεις του Συμβουλίου και πολλών χωρών μελών. Είναι παρόντα νομίζω τώρα και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσαμε πολλά σχετικά με το joint instrument. Εμείς ζητήσαμε και νομική συμβουλή για τον δεσμευτικό χαρακτήρα του joint instrument. Αλλά ιδίω για τις δηλώσεις του Συμβουλίου θα ήθελα να ακούσω από τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου τι λέει η Προεδρία για το νομικό καθεστώς της δήλωσης αυτής. Σε ό,τι αφορά αυτό το κοινό έγγραφο, joint instrument, υπάρχουν κάποια ζητήματα εκεί, για παράδειγμα για τις δημόσιες προμήθειες, για τα περιβαλλοντικά κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιούνται, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης για τα υποχρεωτικά ε, συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων. Οι δηλώσεις σχετικά με το Joint Instrument λένε καθαρά ότι εξαιρούνται τα συστήματα αυτά από την συμφωνία. Και αυτά ε, ανταποκρίνονται στις επιθυμίες μας. Υπάρχουν και άλλα θέματα, γνωρίζετε άλλωστε την θέση μας, που δεν μας ικανοποιούν. Όμως ομολογώ ότι στα δύο θέματα που προανέφερα βλέπουμε κάποια πρόοδο και αυτό είναι καλό. Μένουν όμως κάποια ανοιχτά θέματα. Συνολικά, εγώ νομίζω ότι καλά κάνουμε και συζητούμε πανευρωπαϊκά την εμπορική πολιτική. Ως τώρα ποτέ δεν είχε γίνει. Είναι καλό λοιπόν που βγαίνουν στο φως τα επιχειρήματα αυτά και χαίρομαι που καθένας και καθεμία έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα επιχειρήματά τους και δημόσια, και εγώ πάντως το κάνω αυτό συχνά. Ας μην φοβόμαστε τη συζήτηση αυτή. Είναι καλύτερα να γίνει η συζήτηση αυτή σχετικά με το ποιο θα είναι το μέλλον της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής. Πολλά θέματα έχουν φορτωθεί στην εμπορική πολιτική και θα πρέπει να διεξαχθεί και ένα διάλογο και εδώ στην παρούσα Επιτροπή για το ποια μορφή θα πρέπει να λάβουν οι εμπορικέ συμφωνίε του μέλλοντος, αλλά και για τι διαδικασίε. διότι συμφωνώ και εγώ ότι ήταν ακατάστατη η διαδικασία και δεν θα πρέπει να είναι. Και εμεί ω Επιτροπή ΙΝΤΑ πρέπει να παίξουμε ένα εντονότερο ρόλο. Σωστό. Και εμεί έχουμε και κάποιε προτάσει για το πώ μπορούν να βελτιωθούν οι διαδικασίε, Για παράδειγμα, με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη από την φάση τη χορήγηση τη εντολής και όχι πάντα να προτείνει το περιεχόμενο τη εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το δέχεται το Συμβούλιο και εμεί να μένουμε απ' έξω. Έχουμε λοιπόν κάποιε προτάσει που μπορούμε να κάνουμε, Βεβαίω άλλε πολιτικέ ομάδε έχουν άλλε ιδέε, αλλά επιτέλου α το κάνουμε και πέραν από την εμπορική συμφωνία που έχουμε σήμερα ενώπιόν μα. Εκτός από τα νομικά θέματα, έχω και ερωτήσεις για την δήλωση του Συμβουλίου, ειδικότερα. Διότι υπήρξε και ένα άλλο βελγικό αίτημα, να λεχθεί δηλαδή ότι αν το κεφάλαιο ICS δεν τροποποιηθεί, μπορεί η Προεδρία ή το Συμβούλιο κάποιος άλλος να μου εξηγήσει πώς θα προχωρήσουμε. Τώρα υπογράφηκε η Συμφωνία ΣΕΤΑ. Αν όμως κατανοώ σωστά, η Βελική Συμφωνία λέει ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το κεφάλαιο ICS, δηλαδή της διαιτητικής επίλυσης διαφορών, η ΔΕΜΗ δεν θα υπογράψει τελικά το ε, Βέλγιο. Και τέλος ποιο είναι το χρονοδιαγράμμα για το ε, αίτημα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν θα πω τίποτα για το χρονοδιάγραμμα, ε, διότι και χάσαμε. Αλλά υπήρχε και το θέμα της εμπλοκής των εθνικών κοινοβουλίων. Τα εθνικά κοινοβούλια όμως αυτό σημαίνει μόνο τις εμπορικές επιτροπές της κάθε μια Εθνικής Βουλής, που νομίζω ότι δεν φτάνει. Οι επιτροπές εμπορίου δηλαδή. Ο κ. Πάμπριξ είναι εισηγητή βέβαια. Μήπω μπορεί λοιπόν να διευρυνθεί ώστε να μην έχουμε από κάθε Εθνική Βουλή μονάχα έναν να έρθει εδώ σε ένα γεύμα που θα κρατήσει μια-δύο ώρε και δεν ξέρω καν πόσοι θα λάβουν τον κόπο να έρθουν στι Βρυξέλλε. Χρειαζόμαστε την εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων και πολύ σοβαρά μάλιστα. Και αυτό το έχουν υποσχεθεί και όχι μόνο εδώ, αλλά και σε διάφορες χώρες μέλη. Αλλά όπως είπα, ένας μοναχά εκπρόσωπος από κάθε χώρα μέλος δεν μου φτάνει. Μάλιστα. Τώρα η Τιτσιάνα Μπεγκίνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τόσες φορές που έχω μιλήσει για το ΣΕΤΑ δεν μπορώ παρά να επαναλάβω τα ίδια λόγια. Απλώς θα προσπαθήσω σήμερα να αναπτύξω μια ε, συλλογιστική δεν έφτασαν οι αντιδράσεις των πολιτών, δεν έφτασε το όχι της Βαλονίας, δεν έφτασε καμία προσπάθεια, καμία κυβέρνηση. Τελικά στις 30 Οκτωβρίου υπογράφηκε η ΣΕΤΑ. Ε, τροποποιήθηκε η ψήφος της ε, Βαλονίας από μια συνδυασμένη προσπάθεια της Επιτροπής και των κυβερνήσεων. Το ξέρουμε τόσο ή άλλως ότι ήταν ένας μάταιος αγώνας του Δαβίδ κατά του Γκολιάθ. Αλλά αυτό που βλέπω ότι οι Βαλόνοι για μία φορά ζητούν ε, να αντιδράσουν σε μια ιδιωτική δικαιοσύνη και βρίσκονται ενώπιον ε, κάποιων ε, ε, φιλοδοξιών για απελευθέρωση του εμπορίου που όμως θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της. Είναι σημαντικό το αφήγημα κυρίες και κύριοι αγαπητέ, αγαπητέ Πρόεδρε. Η δημοκρατία στην Ευρώπη είπαν κάποιοι κινδυνεύει γιατί μια μικρή περιφέρεια που σας υπενθυμίσω είναι μεγαλύτερη από ορισμένα κράτη-μέλη ε, τόλμησε να αμφισβητήσει μια ε, διατλαντική συμφωνία. Κυρώνεται, λοιπόν και ακριβώς επειδή κυρώθηκε αυτή η συμφωνία κοινωνία κινδυνεύει η δημοκρατία, γιατί δίνουμε έτσι στις πολυεθνικές το δικαίωμα να μας προσαγάγουν σε δίκη, γιατί τους δίνουμε το δικαίωμα να παρεμβαίνουν στην ομοθεσία μας, γιατί τα δικαιώματα τα υπάγουμε στον όρο τη οικονομική ανάπτυξη. Και ξέρετε γιατί κινδυνεύει η δημοκρατία, γιατί ακριβώ αυτό έχει συμβεί πάντοτε στην Ευρώπη. Όταν δηλαδή κάποιο εκδηλώνει την αντίθεσή του σε, μια, σε ένα εγχείρημα, τον βάζουμε να ξαναψηφίζει μέχρι να αλλάξει γνώμη. Και τελικά μετατρέπουμε την ψηφοφορία σε έναν ε, ε, σε έναν τρόπο να δείξουμε την άγνοια του κόσμου. Ε, το είδαμε το αποτέλεσμα του Brexit, είδαμε το αποτέλεσμα του, των εκλογών στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ο, ο άκρος νεοφιλελευθερισμός είναι αυτός το οποίο, ο οποίος δίνει φωνή σε αυτόν ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ε, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο σοφοί, πιο θαραλέοι, να γίνει μια συζήτηση σοβαρή. Και θέλω να πιστεύω ότι θα δείξουμε και το θάρρος να λέμε όχι σε συμφωνίες ή τουλάχιστον να λέμε το ναι σε συμφωνίες πιο δίκαιες. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει εξ ονόματος του ΙΕΝΕΦ. Ο κ. Σομπερμάγερ ή... Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με τη ΣΕΤΑ θα επιβάλλετε στους Ευρωπαίους ένα πολύ αυστηρό καθεστώς και θα σας το περιγράψω σύντομα. Με την εξαίρεση κάποιων ε, λίγων υπηρεσιών, η δημόσιος τομέα θα μπει στον εμπορικό τομέα. Θα χρησιμοποιήσετε όλα τα κόλπα του ΠΟΕ για να εμποδίσετε στην πράξη τα κράτη να προστατεύσουν νόμιμα και θεμητά τους πολίτες τους με τους γεωργούς. Εδώ βάλατε, ισοπεδώσατε τη γεωργία της Γαλλίας με το φιλελεύθερο σας ε, πρόσωπο και την αφήσατε ε, ακάλυπτη απέναντι σε, μια έναν εξαιρετικά αθέμητο ανταγωνισμό. Με τους ε, Καναδούς ε, γεωργούς. Το κόστος τους μάλιστα θα είναι 35% χαμηλότερο στον Καναδά χάρη στην εντατική χρήση ε, των αντιβιωτικών. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ακόμα και αυτοί που ήθελαν θα προστατευθούν, δεν θα προστατευθούν. 42 επιχειρήσεις μόνο στη Γαλλία θα προστατευθούν, αλλά θα είναι πολύ περιορισμένη η πρακτική αυτή. Τώρα, για τις πολυεθνικές και τη δυνατότητα ε, δίκης κατά των κρατών μας, αυτό το καλύψατε, το καμουφλάρατε με αυτό το ε, υποτιθέμενο σύστημα για τις επενδύσεις, ε, όμως οι δικαστές θα πληρώνονται από τις ίδιες, πολλές φορές από τις ίδιες τις ε, πολυεθνικές. Τέλος, για τα εθνικά κοινοβούλια, ε, κάντε λες και δεν μετράνε. Αν πούν όχι, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα το κάνουν. Σταματήστε, πάψτε, η δική μας βούληση είναι ανώτερη λέτε. Έχω μια ερώτηση. Ο Ντόναλτ Τραμπ, που είναι πρόεδρος της πρώτης παγκόσμιας δύναμης, έχει υποσχεθεί πως οι ΗΠΑ θα φυγούν από το ΠΟΕ και θα γίνουν προστατευτική δύναμη. Ε, εσείς θέλετε να παραμείνετε δογματικά φιλελεύθεροι ενώ οι άλλες δυνάμεις υιοθετούν πολιτική ε, που είναι τελείως αντίθετη με τη δική σας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κασπάρη. Ευχαριστώ αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι και περισσότεροι ανησυχούν. Τα ακούμε και εμείς αυτά. Τι γίνεται με την παγκοσμιοποίηση, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό χωρών όπως Κίνα, Ινδία, Βραζιλία. Βλέπουμε και τους χαλιβουργούς σήμερα που διαμαρτύρονται και διαδηλώνουν. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά. Από την άλλη μεριά ωστόσο Ήδη 14% των θέσεων απασχολήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτώνται από τις εξαγωγές. Για κάθε δισεκατομμύριο 14.000 εξαγωγών, δηλαδή αξίας εξαγωγών σε ευρώ, 14.000 θέσεις εξαρτώνται από αυτά. Αρχίζουν τώρα, είτε λοιπόν θα συμμετάσχουμε στην προσπάθεια αυτή, αλλά τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδιαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση. Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν το διεθνές εμπόριο. Δεν... Πώς θα εξασφαλίσουμε τα ε, ε, πρότυπά μας περιβαλλοντικά και άλλα, την πολιτιστική μας ποικιλία, το πολιτιστικό τοπίο, πώς θα βελτιώσουμε όχι μονάχα για τους μεγάλους αλλά και για τις πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τις δυνατότητες εξαγωγών ώστε και αυτές να μπορέσουν με τη σειρά τους να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις απασχολήσεως. Πώς θα εξασφαλίσουμε στην εξαγωγική μας βιομηχανία πρόσβαση στις αγορές εάν όλο και περισσότερες χώρες λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα. Πώς θα διασφαλίσουμε ώστε και πολλές και πολλοί προμηθευτές, δηλαδή πολλές εταιρείες μα, οι οποίε δεν εξάγουν οι ίδιες μεν, αλλά προμηθεύουν τα ειδικά σε αυτές οι οποίες εξάγουν. Πώς θα εξασφαλίσουμε λοιπόν και αυτή την επιχείρηση και όλο το προμηθευτικό τομέα. Πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την πώληση των προϊόντων μας, την ε, προστασία των γεωγραφικών μας προελεύσεων. Σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, ωστόσο, η ΣΕΤΑ δίνει πολύ ξεκάθαρες και καλές απαντήσεις. Πέντε χρόνια διήρκησαν οι διαπραγματεύσεις και ούτε περνούμε την ε, συμφωνία αυτή με ταχύτατες διαδικασίες όπως προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε ορισμένοι συνάδελφοι. Εδώ και δύο χρόνια εξετάζουμε την συμφωνία. Έγιναν βελτιώσεις, έγιναν νέες διαπραγματεύσεις για θέματα των διαιτητικών επιλύσεων διαφορών, για παράδειγμα ακόμα και τις τελευταίες εβδομάδες και εύχομαι πραγματικά να δώσουμε περισσότερη σημασία και να διαφημίσουμε ακόμη περισσότερο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν εμπλεκόμενο και τα 7 χρόνια. Πάντοτε εξαγάγαμε τακτική συνεννόηση και με, τις, ε, ε, και με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με τις κυβερνήσεις και μάλιστα και με θεσμικό τρόπο θεσμοποιήσαμε τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια και όχι μόνο με βουλευτές αλλά ακόμα μέχρι και με τους συνεργάτες και στις 29 Νοεμβρίου δεν θα έρθει ένας βουλευτής μονάχα από κάθε Εθνική Βουλή. Οι προσκλήσεις απευθύνθηκαν στους επικεφαλής, στους προέδρους των επιτροπών. Βεβαίω μπορούν να έλθουν όλοι οι βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια που επιθυμούν να συζητήσουν το θέμα. Το θέμα της Γεωργίας. Εκεί η αλήθεια είναι ότι ε, ε, ε, λόγω της ΣΕΤΑ δεν πρόκειται να έλθει, δεν απειλείται να έλθει ορμονούχο κρέας στην Ευρώπη. Με τη ΣΕΤΑ το αποφεύγουμε αντιθέτως αυτό. Μέσα, μέσω της ΣΕΤΑ εξασφαλίσουμε ότι το ορμονούχο κρέας παραμένει απ' έξω. Δηλαδή για τις εξαγωγές του κρέατος οι Καναδοί θα παράγουν σύμφωνα με τα δικά μας πρότυπα. Και μάλιστα είπαν οι Καναδοί ότι θα το τροποποιήσουμε, μάλιστα λένε, ολόκληρη την παραγωγή μα και θα χρησιμοποιήσουμε τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα, όχι μόνο για να μπορούμε να πολλούμε το κρέα στην Ευρώπη, αλλά θα χρησιμοποιήσουν τα υψηλότερα αυτά πρότυπα και για τον ίδιο τον Καναδά. Να έχουν καλύτερο κρέα για να μπορούν να πολλούν και στου ίδιου του Καναδού κρέα χωρί ορμόνε. Άρα στην ουσία εξάγουμε τα πρότυπα και τι προδιαγραφέ μα και για τι γεωγραφικέ προελεύσει δεν παραχωρούμε τίποτε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορέσαμε να ε, προστατεύσουμε και τις 41 γεωγραφικές προελεύσεις ή τις 1000 συνολικά ευρωπαϊκές γεωγραφικές προελεύσεις στον το ίδιο τον Καναδά. Όμως βάλαμε επιτέλους ένα φρένο ότι να δεχθούν επιτέλους ότι υπάρχουν και στις ΗΠΑ και στη Βόρεια Αμερική δηλαδή συνολικότερα, υπάρχει κάτι που λέγεται γεωγραφική προέλευση. Διότι μέχρι τώρα δεν προστατεύεται καμία απολύτω γεωγραφική προέλευση στον Καναδά ή στη Βόρεια Αμερική. Και εάν επανέλθουμε στην ΣΕΤΑ και την αναπτύξουμε ξανά μετά από 10-15 χρόνια, θα πούμε τότε δεν θέλουμε μόνο 140 γεωγραφικέ προελεύσει, αλλά θέλουμε 200-300 που να προστατεύονται. Εκεί λοιπόν επίση η ΣΕΤΑ δεν αποτελεί κίνδυνο όπω του και ισχυρίστηκαν μόλι πριν, Αντίθετα, προστατεύει τους γεωργούς μας στον όλο και ισχυρότερο ανταγωνισμό. Και επίσης για, τις, ε, για την ε, παροχή κοινοτικών αγαθών στις επίπεδο των κοινοτήτων, δηλαδή πάλι εκεί δεν ε, πέφτουν οι προστασίες αντιθέτως. Ελπίζω μάλιστα ότι θα μπορέσει να ψηφιστεί η συμφωνία ήδη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέτο, μέχρι τέλο του έτου, ώστε να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου. Ελπίζω και οι χώρε μέλη να κυρώσουν την καλή αυτή συμφωνία όμως προπάντων χρειάζεται μια έντιμη συζήτηση. Μην, μην ε, φόβους που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την προκείμενη συμφωνία. Η κατάσταση που είδαμε τις τελευταίες ε, εβδομάδες της συζητήσεως ήταν αξιοδάκριτη. Πρέπει κάθε επίπεδο να παίξει τον ρόλο τους. Όπως οι τοπικές κοινότητες ενοχλούνται όταν αναπηγνιόμαστε εμείς, έτσι και εμείς πρέπει να πούμε καθαρά ότι προσέξτε, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις λαμβάνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό θα πρέπει να παραμείνει στόχος μας, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει και στο μέλλον να συνδιαμορφώνει την παγκοσμιοποίηση, διότι αυτό το χρωστάμε τελικά στους ανθρώπους στην Ευρώπη. Dankeschön. Und nun ist Maria Arena dran. Ευχαριστώ, κυρία ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω εξ αρχή στον κύριο Κασπαρή ότι το να γίνεται τίμια συζήτηση δεν σημαίνει ότι όσοι επικρίνουν πρέπει να παίρνουν την ετικέτα της Βόρειας Κορέας ή να βάζουμε λόγια στο στόμα του Επιτρόπου Ότιγκερ. Η σωστή συζήτηση δεν σημαίνει να προσβάλλουμε τους άλλους. Ελπίζω, ε, θα ήθελα μάλλον η διόρθωση να εφαρμοστεί και από τις δύο πλευρές και όχι μόνο από τη μία. Δεύτερον, φυσικά και συμφωνούμε για το διεθνές εμπόριο. Χρειάζεται διεθνές εμπόριο και υπάρχει και πρέπει και να υπάρχουν και κανόνες μάλιστα. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα στους κανόνες αυτούς βλέπουμε ότι δεν είναι όλοι οι κανόνες αυτοί εγγυημένοι. Και όταν είδαμε Βέλγους και πιο συγκεκριμένα Βαλώνους να θέτουν ερωτήματα ε, εδώ και δύο χρόνια για αυτό στους κανόνες και να μην παίρνουν απαντήσεις επειδή θέσαμε τις ίδιες ερωτήσεις εδώ, στο Κοινοβούλιο εδώ και δύο χρόνια και δεν πήραμε απαντήσεις σε κάποια στιγμή θα πρέπει να λάβουμε κάποια θέση και ίσως και να είναι κάπως ισχυρές ναι, οι θέσεις αυτές αλλά λήφθησαν και επιπλέον θέλω να πω ότι αν δεν είχε υπάρξει αυτή η αβεβαιότητα σε σχέση με την, το μεικτό χαρακτήρα αυτής της ε, συμφωνίας, ε, αβεβαιότητα ε, που δεν αμβλήθηκε ούτε από τους Βαλώνους, ούτε από τους ε, ε, Βέλγους, ούτε από κάποιο άλλο μικρό κράτος, αλλά, μικτός χαρακτήρας που ζητήθηκε στο Συμβούλιο από τη Γαλλία και από τη Γερμανία και όπου η Κομισιόν απάντησε σε πολιτικό επίπεδο και είπε εμείς θεωρούμε αυτή τη συμφωνία μεικτή. Από τη στιγμή που λήφθη τέτοια απόφαση αυτή, απόφαση δηλαδή να είναι μεικτή αυτή η συμφωνία, και πολύ θα ήθελα να ήταν απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί τότε δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από κανέναν. Σήμερα έχουμε μια πολιτική απόφαση λοιπόν για το μειχτό χαρακτήρα και κατηγορείται ένα κράτος μέλος επειδή έκανε τη δουλειά του. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε αρμοδιότητες, τις ασκούμε στο κομμάτι που μας αφορά. Λοιπόν, ε, θέλω να πω εδώ ότι εφόσον αυτή εδώ η Δημοκρατική Συνέλευση είναι δημοκρατική συνέλευση και πρέπει να τη σεβαστούμε. Τα κράτη-μέλη όταν τους δίνουν ε, την αρμοδιότητα ε, και αυτά είναι δημοκρατικά. Όσο και η δική μας συνέλευση. Γι' αυτό θα πρέπει να αποσαφινιστούν τα πράγματα όσον αφορά το μειχτό χαρακτήρα και να αποφευχθεί ο ερασιτεχνισμός που ζήσαμε μέχρι σήμερα ανάμεσα στην Κομισιόν και το Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω να περιμένουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ψήν να ψηφίσουμε για αυτή την συμφωνία, γιατί δεν γνωρίζουμε ε, επί ποιου θα πράγματα θα ψηφίσουμε. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αποκλειστική μας αρμοδιότητα ως Ευρωκοινοβούλιο και τι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Άρα λοιπόν θα ψηφίσουμε κάτι με, που θα αρχίσει να ισχύει προσωρινά, αλλά για το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώ τι θα αρχίσει να ισχύει προσωρινά. Και ακόμα πιο άλλη μια δυσκολία είναι ακριβώς αυτές οι ερμηνείες, οι δηλώσεις μάλλον ερμηνευτικέ, που είναι δεσμευτικές, είναι μέσα, είναι εργαλεία, είναι δηλώσεις με το σύνολο των φορέων ή μονιμερείς των κρατών μελών δηλώσεις. Τρία διαφορετικά νομικά καθεστώτα που μας οδηγούν στο να μην ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα θα ψηφίσουμε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με τον Καναδά όπου υπάρχει το ICS, το σύστημα ε, δικαστηρίου για τις επενδύσεις. Το Βέλγιο όμω είπε, εμεί δεν πρόκειται να κυρώσουμε τη συμφωνία από τη στιγμή που δεν έχει τροποποιηθεί το ICS. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ICS, όπω αυτή τη στιγμή είναι επιτάπητο. Ποιο ICS θα έχουμε. Εδώ θα ψηφίσουμε για ένα ICS, το οποίο όμω μάλλον με τη μορφή που μας έχει παρουσιαστεί, ξέρουμε πως δεν θα επικυρωθεί, δεν θα κυρωθεί, γιατί ένα κράτος μάλλον δεν θα το κυρώσει αυτό και άρα δεν πρόκειται να αρχίσει να ισχύει. Η Κομισιόν μας λέει ότι παίρνω την δέσμευση, αναλαμβάνω τη δέσμευση να το τροποποιήσω, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα τροποποιηθεί. Δηλαδή ψηφίζουμε για ένα ICS ε, ε, εκδοχή Α που θα τροποποιηθεί, δεν ξέρουμε πώς θα, αν θα γίνει δεκτό και παρόλα αυτά θα το ψηφίσουμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Πιστεύω πως πρόκειται για έναν απίστευτο αριστεχνισμό και κύριε Πρόεδρε είπατε πρέπει να τηρήσουμε τη δημοκρατία εδώ. Εφόσον θέλουμε λοιπόν να κάνουμε τη δουλειά μας ως ευρωβουλευτές, και όχι να κατευθυνόμαστε από τις πρωτεύουσέ μας, αλλά τη δική μας δουλειά ως Ευρωβουλευτές, ζητώ να έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συγκεκριμένες και πρακτικές για το τι θα ψηφίσουμε ακριβώς στις επόμενες εβδομάδες. Και ακριβώς τότε θα είμαστε αξιόπιστοι. Άμα δεν ξέρουμε τι ψηφίζουμε, θα μας επιτεθεί ο πληθυσμό που θα πει πιέσατε το πράσινο κουμπί και δεν, χωρίς να ξέρετε καν τι δεχτήκατε ή πατήσατε το κόκκινο κουμπί γιατί δεν ξέρετε καν ε, τι πρέπει να ψήσετε. Σοβαρότητα λοιπόν από πλευρά ε, Συμβουλίου, Κομισιόν και Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάκουλα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ύστερα από αυτές τις δύο καλές και τόσο θυελώδεις παρεμβάσεις των δύο συναδέλφων, τόσο πλούσιες μάλλον. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο πιο φιδωλά. Είδαμε ότι υπάρχουν πολλά, πολλοί αστάθμητοι παραγόντες ως ε, προς την στάση των κρατών μελών στην εμπορική πολιτική. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποια είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία μέχρι τώρα έχουν ε, κοινοποιήσει πρόθεση να απόσχουν ή να δράσουν αντίθετα με τους όρους της Συμφωνίας Εμπορικών Σχέσεων. Γιατί νομίζω ότι όλες οι κυβερνήσει πιστεύουν, συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε ε, μια εμπορική πολιτική που θα στηρίσει στους ώμους των 28 κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό και ότι είναι πολύ πιο ε, συμφέρουσα αυτή η στάση παρά το να προσπαθεί το κάθε κράτος μόνο του να συναπτύει εμπορικέ σχέσεις. Γιατί στη χώρα μου και οι πιο σκληροί ακόμα κομμουνιστές, οι πιο σκληροί ε, δεξιοί λένε όχι θα φροντίσουμε να προχωρήσει και η ΣΕΤΑ να υλοποιηθεί για να φέρει νέα δουλειά στα ναυπηγεία μας. Άρα βλέπω ότι όλες οι δυνάμεις τίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Ήταν ενδιαφέρουσα για μένα η παρατήρηση αυτή σε σχέση με την ΣΕΤΑ, γιατί βλέπω και μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι οποίες ε, είναι πολύ δραστήριες ε, και στα κοινωνικά μέσα κτλ. να μιλούν αλλά η πολιτική, το πολιτικό φάσμα όλο από την δεξιά μέχρι την αριστερά ε, είναι σύμφωνο. Άρα δεν υπάρχει θέμα τυχόν πολιτικών στην υπόθεση αυτή. Και μια και ήρθε ο λόγος με τύχη. Θυμήθηκα τον ε, μελλοντικό πρόεδρο των ΗΠΑ, τον ε, Τραμπ. Ίσως να μην πρέπει να παίρνουμε στα, καταγράμματα λόγια του. Πολλές φορές λέγονται πράγματα τα οποία μετά δεν τηρούνται ή σημαίνουν κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλοι στην Επιτροπή μας συμφωνούμε πως πρέπει να υλοποιηθεί η ΣΕΤΑ. Και βέβαια, καλό είναι να δούμε και στη συνέχεια η νέα ε, κυβέρνηση των Πολιτειών τι στάση θα τηρήσει. Ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις βλέπουμε να ε, τίθεται ένα αμφιβόλο η κύρωση της ΣΕΤΑ και ίσως θα έπρεπε να αλλάξουμε λίγο τη διαδικασία και να φροντίσουμε στο μέλλον η κύρωση να περνάει μόνο μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια δεν ξέρω τι ε, ετοιμιγορία θα εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά θα είναι χρήσιμο να το κοιτάξουμε αυτό. Και έτσι να είναι σε θέση να εξασφαλίσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται και να εγκρίνει ως σύνολο αυτές τις συμφωνίες. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω ότι το χειρότερο δυνατό να περάσει η κύρωση από όλα τα κράτη ώστε να υλοποιηθεί ε, η ΣΕΤΑ το ταχύτερο. Και πιστεύω ότι είναι πάντα καλό να γίνεται ειλικρινή συζήτηση. Αλλά ταυτόχρονα να προσέχουμε και τις παρεξηγήσεις ή παρερμηνίες των λόγων μας σε τέτοιου είδους ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις. Εμείς ως βουλευτές οφείλουμε να αντιλαμβανόμεθα το πραγματικό νόημα των λόγων, να εξαρτήτως των προθέσεων εκείνου που, τις, ε, ε, που τους εκφωνεί ή που τα ξεστομίζει. Και πάνω απ' όλα να εργαζόμαστε για το καλό των περιφερειών μας. Σας ευχαριστώ. Εμμανουέλ Μαουρέλ. Ευχαριστώ. Πολύ θετικό το ότι ε, ανέλαβε να διεξαγάγει τη δημόσια συζήτηση η κοινή γνώμη για τη ΣΕΤΑ. Νομίζω ότι αυτό και για εμάς τους βουλευτές που συζητάμε τόσο καιρό το διεθνές εμπόριο είναι πολύ θετικό το να βλέπουμε δηλαδή ότι το θέμα αυτό εγγράφεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινή νόμης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι συναρπάζει τον κόσμο τόσο. Γιατί κατάλαβε ο κόσμος ότι υπάρχουν και οι κίνδυνοι, υπάρχουν και οι ευκαιρίες. Είναι καλό το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση. όλοι μιλάνε για τον Ντόναλτ Τραμπ αλλά στο επίκεντρο της ε, προεκλογικής του εκστρατείας ήταν ακριβώς το θέμα των ελεύθερων συναλλαγών και μεγάλο κομμάτι της συζήτηση ε, και του δημόσιου διαλόγου στις ΗΠΑ, όχι μόνο μεταξύ ε, ρεπουμπλικανών αλλά και μεταξύ δημοκρατικών, ήταν το τι συνέπειες θα έχει η ναύτα και αν θα συνεχίσει να τηρείται. Και ξέρουμε ότι αυτό επικράτησε στη συζήτηση με τα γνωστά αποτελέσματα βεβαίως από την εφαρμογή. δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αυτή τη συζήτηση. Και δεν καταλαβαίνω αυτούς ε, που λένε ότι α, η, αντίθε, η, οι πολέμοι των συμφωνιών δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να απλοποιούν ε, τους όρους της συζήτησης, που όντως συμβαίνει πολλές φορές, αλλά δεν μπορούμε να εξαντλούμε συζήτηση αυτό, ούτε βέβαια και την κατηγορία ότι αν είσαστε κατά της συμφωνίας θέλετε σύστημα Βόρειας Κορέας και Σοβιετικής Ένωσης. Και επίσης όταν γίνεται λόγος για την ε, ε Βαλόνια, θα απαντήσω ότι όταν ένα πολύ πολύ μικρό κρατήδιο, όπως το Λουξεμβούργο παρεμποδίζει οποιαδήποτε εξέλιξη σχέση με τα φορολογικά, Κανεί δεν μιλάει και δεν το ακούμε καν ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όταν μια περιφέρεια που δεν είναι και τόσο μικρή σε τελευταία ανάλυση, είναι μεγαλύτερη από κράτη, μέλη, ε, παρεμποδίζει γιατί έχει κάποια ερωτηματικά και θέλει απαντήσεις μια συμφωνία εμπορίου, όλοι αμέσως αρχίζουν να ξελαψουρίζουν. Ο Πολ Μανιέτο, πρόεδρο τη περιφέρεια, έδωσε απαντήσει, οι οποίε είναι έγκυρε για κάθε περιοχή Τη Ευρώπης και δεν ξέρω ίσως τι συμβαίνει γιατί στην ε, Φινλανδία ή στη Γερμανία αλλά σας διαβεβαιώ ότι αν γινόταν αντίστοιχο δημοψήφισμα στη Γαλλία γιατί αυτή τη γνωρίζω καλά θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Επομένω, τα ερωτηματικά των βαλώνων βουλευτών είναι έγκυρα και εκπροσωπούν όλου του πολίτε. Επίση, εάν κοιτάξουμε προσοχή το κείμενο, πολλά είναι τα εκρεμή ζητήματα το πρώτο εκρεμέ ζήτημα και μάλιστα ποτέ δεν δόθηκε απάντηση από την Επιτροπή από το Συμβούλιο, από τι Υπηρεσίε του Κοινοβουλίου, είναι τι προβλέπεται να έχουμε ω οικονομικό όφελος. Γιατί κάθε οικονομική συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να φέρνει οικονομικό κέρδο, αλλά δεν είναι αρκετά φιλόδοξη από ό,τι βλέπουμε συγκεκριμένη. Καλή η ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών για την ανάπτυξη, την απασχόληση, αλλά σε πραγματικό οικονομικό κέρδο δεν βλέπω τίποτε το σαφέ. Πρώτον. Δεύτερον, και για να επανέλθω στα όσα είπε ο κύριος Κασπάρη, ε, και όλα αυτά τα λυρικά και ε, ε, συγκινητικά για τη γεωργία της Ευρώπης. Μα, κοιτάξτε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα έρθει ένα επιπλέον ποσ... μια επιπλέον ποσόστοση βόηου και χείριου κρέατο που θα έρθει στην Ευρώπη. Λέτε ότι είναι υπολογισμένο. Ναι, αλλά αυτό είχε υπολογιστεί με βάση και την παρουσία τη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μετά τον Brexit βρισκόμαστε σε μια ιδιάζουσα κατάσταση όπου θα πρέπει να, να προσαρμοστούν αυτές οι ποσοστώσει. οι τόνοι κρέατο βοήου και χειρίου που πρέπει να εισαχθούν. Τρίτο ερωτηματικό εκρεμές αμφιβολίες πολλές σε σχέση με τις ερμηνείες, δηλώσεις, κοινέ δηλώσεις, διακηρύξεις που βρίσκονται πλέον επιτάπητος. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Πρώτον, συμβατότητα μεταξύ του συστήματος διαιτησίας και του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεύτερον, ζήτημα συνταγματικότητας ορισμένων εκτών διατάξεων. Υπάρχουν πολλοί συνταγματολόγοι που έχουν εκδώσει ε, μελέτη στη Γαλλία που μας λένε ότι είναι αντισυνταγματικά ορισμένα σχετικά με τη ε, ε, ρύθμιση, με τους κανόνες. Ζητήματα νομοποίησης του μηχανισμού προσωρινής εφαρμογής. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Η Γερμανία έχει εξασφαλίσει ένα μηχανισμό του opt-out σε σχέση με την προσωρινή εφαρμογή. Το Βέλγιο επίσης. Τα άλλα κράτη μπορούν ή δεν μπορούν. Δεν έχω καταλάβει τι ισχύει. Μπορεί να είμαι και ανόητο, τι να πω, αλλά πάντω να έχω καταλάβει. Ε, για δε τις δηλώσεις επιτροπής προβλέπεται η αρχή της πρόληψης. αλλά στο κοινό ερμηνευτικό ε, κείμενο που εκδόθηκε μαζί με τον Καναδά δεν προβλέπεται η αρχή της πρόληψης την οποία ξέρουμε ότι στον ΠΟΕ ε, καταπολεμούν με τα μανία οι και ο Καναδάς Άρα είναι πολλά τα εκκρεμή ζητήματα. Αυτά δεν είναι ούτε φαντασιώσεις, ούτε ε, προσδοκίες να γίνουμε Βόρεια Κορέα είναι απορίες πραγματικές και μάλιστα νομικού περιεχομένου. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί ο χρόνος να δοθούν οι απαντήσεις, να γίνει η συζήτηση και, εν πάση περιπτώσει, ας εκδηλώσουμε και την ικανοποίησή μας που τους ενδιαφέρει τους πολίτες της Ευρώπης ένα τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τον Άγιο Πολίτη αίσθημα ότι τα πάντα γίνονται εν και παραβίστο. Ας γίνει αυτή η συζήτηση και ας τη συνεχίσουμε εμείς. Είναι συναρπαστική. David Martin. Ο κύριος David Μάρτιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ξέρω αν όντως είναι παρόν το Συμβούλιο. Βλέπω ότι κάποιοι κάθονται στα καθίσματα για να απαντήσουν. Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνονται στο Συμβούλιο και όχι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι που ο Μάουρο είναι παρόν πάλι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε μας έχει ενημερώσει. Σωστά είπατε όμως και εσείς αρχικά ότι το Συμβούλιο δεν έχει τηρήσει τις συνθήκες. Και αντιθέτως από αυτά που είπε ο Μαουρίσιο, νομίζω ότι πολύ καλά έκανε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και αναμίχθηκε στην συζήτηση. Διότι αν δεν είχε υπάρξει και αυτή η παρέμβαση, τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου θα είχαν εντελώς καταπατηθεί και τουλάχιστον με τη στάση του κατέστησε σαφές και στους άλλους της και στους Καναδούς ότι το Κοινοβούλιο παίζει ένα ρόλο. Έτσι λοιπόν οι ανησυχίες μου αναφέρονται κυρίως στη στάση του Συμβουλίου. Ο Μανουέλ είπε Γερμανοί, Πολωνοί και Βέλγοι που έχουν ζητήσει εξαίρεση από την προσωρινή εφαρμογή. Τι σημαίνουν και αυτή η προσωρινή εφαρμογή τι σημαίνει. Μιλούμε υποτίθεται για αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, αυτές οι εξαιρέσεις είναι ασυμβίβαστες με την ε, συνθήκη. Πώς μπορεί κάποιο κοινοβούλιο να εξαιρέσει από την εφαρμογή τμήμα της συνθήκης. Κάτι το οποίο υποσκέπτει και την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Και συμφωνώ με τη Μαρία Ρένα ότι η δεύτερη βαλόνη τους δόθηκε η δυνατότητα να αμφισβητήσουν την συμφωνία. Δεν θα έπρεπε ωστόσο να έχουν φτάσει σε αυτή τη θέση. Αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τη συνθήκη Λισαβόνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την αρμοδιότητα να κυρώσει. Και όπω είπαν και ορισμένοι, υπάρχει κάποια σύγχυση. Τι πάει να πει αποκλειστική αρμοδιότητα, αυτό μας απασχολεί για την βιώσιμη ανάπτυξη που λέει η προσωρινή εφαρμογή των ε, κεφαλαίων 22, 23 και 24 σέβονται την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών. Μα ποια είναι η κατανομή των αρμοδιοτήτων στο κεφάλαιο αυτό. ιστορικά τα κεφάλαια της ε, βιώσιμης ανάπτυξης θεωρούνται αποκλειστική αρμοδιότητα. Πάμε να αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού, λοιπόν, εδώ. Είναι χρήσιμο, λοιπόν, να μας δοθούν οι σχετικές εξηγήσεις. Και πέραν από τη ΣΕΤΑ, η βελγική διακήρυξη για το ICS, τι σημαίνει ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι να έχουμε επιτάπητος νέα μορφή ICS πριν να συζητήσουμε τις συμφωνίες με το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη ή θα θεωρήσουμε ότι θα μπουν σε ένα διαφορετικό κουτί και θα προχωρήσουμε και χωρίς αυτές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Να πούμε ότι μία μορφή ICS μπορεί να ισχύει για μία ε, συμφωνία και άλλη για άλλες. Χρειαζόμαστε και εδώ κάποιο ξεκαθάρισμα. Επίσης κάποιος μίλησε για την αγροτική διακήρυξη. Τι σημαίνει πάλι αυτό. Πού βρίσκεται το κατόφλιο και ποιο κατόφλιο θα υπερπηδηθεί για να αναλάβουμε δράση διαφύλαξης, αφού δεν υπάρχει ρήτρα διαφύλαξης με στη συνθήκη. Είμαι βέβαιο ότι ο Μάουρο θα προσπαθήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει ορισμένε από τις ερωτήσεις αυτές, όμως το Συμβούλιο θα έπρεπε κανονικά να είναι παρόν και να απαντήσει. Υποψιάζομαι ότι οι παρόντες εκπροσωποί του δεν θα μπορέσουν να απαντήσουν. Ελπίζω να μπορέσουν, αλλά χρειαζόμαστε κάποιον που να μπορέσει να απαντήσει από πλευρά Συμβουλίου με κάποια αυθεντία. Ευχαριστώ κύριε Σπρούστ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι, όπως ε, και άλλοι από την ομάδα μου, που αυτή η υπογραφή ε, ε, έγινε τόσο λόγω της δουλειά, τόσο δύσκολη ήταν και σημαντική η δουλειά του εδώ, αλλά και του Συμβουλίου και της Κομισιόν ε, εδώ και τόσα χρόνια και έπειτα ήταν και θέμα αξιοπιστίας ε, γιατί όταν ορίζονται οι κανόνες πριν από 5-6 χρόνια με κόκκινε γραμμές και γενικά υπάρχει ικανοποίηση για αυτές τις κόκκινε γραμμές δεν μπορώ να καταλάβω πώ θα μπορούσαμε να καταψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία που για μένα μετά από ανάλυση και θα επανέλθω, είναι μια συμφωνία ε, όπου τα δύο μέρη βγαίνουν κερδισμένα. Θα πρέπει ωστόσο να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις όταν βλέπουμε τη στάση των μέρων και των δε. Το πρώτο ερώτημα είναι και συμμερίζομαι την θέση σας κύριε Πρόεδρε, ότι δηλαδή εδώ έχει εντύπωση ότι το Κοινοβούλιο αφήθηκε, αφήθηκε κατά μέρο. Γιατί από τη στιγμή που ίσως ήταν μια συμφωνία μεικτή, αυτό ίσως να ήταν λάθος. Μήπως αυτό είναι συνέπεια ε, αυτού ε, και έπειτα με την Κομισιόν ε, φαίνεται να είναι ε, για θέματα διαφάνειας. Θα ήταν καλό να συνδέονται όλο και περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια σε αυτές τις συμφωνίες. Αλλά τότε πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Ε, θα πρέπει να έχουμε το θάρρος. Ο κανόνας της ομοφωνίας είναι σωστός ή μήπως θα πρέπει να περάσουμε σε κανόνες που στόχο θα έχουν να βρεθεί μια ειδική πλειοψηφία ή εξόχως ειδική πλειοψηφία για να μην βρισκόμαστε σε μια τέτοια δύσκολη θέση όπου μια περιφέρεια τριών εκατομμυρίων μπορεί να σταματήσει το μέλλον 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων γιατί όντως εκεί ε, λείπει κάτι. Α πούμε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Να αλλάξουν οι κανόνε. Και έπειτα, εμένα μου αρέσει η συνοχή. Δηλαδή, όντως ότι βγαίνει προς τα έξω στο ευρύ κοινό αυτό το θέμα είναι σημαντικό να δούμε αν θα είναι τόσο ευαίσθητη με τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Διαπιστώνουμε σήμερα ότι το ΣΕΤΑ ή το ΤΑΦΤΑ είναι πιο σημαντικά και ίσως να υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα σε κάποιες μικιό που ασχολούνται ε, με αυτές τις ε, συμφωνίες. Εγώ λοιπόν ε, αγαπώ την συνοχή. Δεν μου αρέσουν οι αναλήθειες ή τα οράματα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν είχε πάει στο, Κοινοβούλιο της Βαλονίας, η κυρία Μάλστρομ είχε πάει, η μιλήσει για δύο ώρες εκεί. Γιατί λοιπόν τότε περίμεναν μέχρι τελευταία στιγμή για να θέσουν αυτά τα ερωτήματα. Στη διάρκεια αυτή τη διάσκεψη δεν υπήρξε, δεν υποβλήθηκε καμιά ερώτηση και υπήρχαν και έγγραφα στου διάφορου τομεί δραστηριότητα. Και αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι ο κύριο Μανιέτ έθεσε διάφορα ερωτήματα ή ανέφερε ανησυχίε. Αυτό είναι απόλυτα θεμητό. Αλλά για 90% οι απαντήσει υπήρχαν μέσα στι 1500 σελίδε τη έκθεση. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Και για πρώτη φορά θα πρέπει να χαιρετήσουμε την εργασία τη Κομισιόν που έκανε ένα σημείωμα που ήταν η πολιτική ερμηνεία, η επεξηγηματική για μια τεχνική σημείωση. Και για πάλι και πάλι, και για να απαντήσω στον συνάδελφο Εμμανουέλ Μορέλα όπου συμφωνώ και εγώ οι Γάλλοι Γεωργοί ήρθαν και μας είδαν και όταν ακούμε και τον κύριο Μαζό, ναι, θα πρέπει να ξαναδιαβάσει την έκθεσή του, γιατί άμα, όταν μιλάει για βόλιο ή για χείριο κρέας, ξέρετε και ο κύριος ε, Κασπαρίτη επανέλαβε, δεν δίνεται δυνατότητα εισαγωγής ε, ε, κρέατος με ορμόνες και οι Καναδοί για να μπορέσουν να εξάγουν κρέας εδώ σε εμά θα πρέπει να ξαναδούν ολόκληρη την αλυσίδα επενδύσεών τους και ε, εκτροφής των ζώων του. Δεν θα γίνει αυτό από την μια μέρα στην άλλη. Αλλά για το βόη έχεις δίκιο. Ε, το θέσαμε την ερώτηση και εγώ πήρα απάντηση. Ανάμεσα στο 13 και το 15 0%, 0% του κρέατος, είτε νοπού, είτε κατεψυγμένου, ε, είτε ε, απλώς ψυγμένου δεν μπήκε από την ε, Βρετανία. Και αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από την αρμόδια γαλλική αρχή. Ναι, να θέτουμε ερωτήσεις, ναι, αλλά να φοβόμαστε φαντάσματα, όχι. Ναι, συζήτηση να γίνει, εννοείται. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει για τη ΣΕΤΑ. Το συζητήσαμε και χτες σε σχέση με αυτή την ημερίδα για την εμπορική πολιτική. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι κατά των πάντων ε, χειραγωγούν την επικοινωνία. Θα πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια στην επικοινωνία, να ενημερώσουμε. Και εδώ θα πρέπει να έχουμε καλύτερη επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια, με τις διάφορες ενώσεις, με τις τομεακές οργανώσεις, για να μπορούμε καλύτερα να επικοινωνούμε. Και έχω βαρεθεί που ορισμένοι θύνοντες πολιτικοί, που δεν έχουν παρά μόνο το όνομα υπεύθυνοι, οι ε, μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι αν αποτύχει μια εμπορική συμφωνία η κατάσταση θα ήταν έκτακτη. Γιατί πιστεύετε πως σήμερα αν δεν συνυπογράφαμε την ΣΕΤΑ οι γεωργοί μας σήμερα προστατεύονται. Κανένας δεν προστατεύεται. Ναι, μπορεί να λέει πως έχουμε μόνο 42. 42 οι οποίε κινδύνευαν, δηλαδή που έφτιαχναν προϊόντα όπου υπήρχε πλαστό προϊόν στον Καναδά, ή προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να εξαγωγθούν. Δεν συγχρησιμεύει σε τίποτα να προστατεύσουμε τις 1.400 ονομασίες προέλευσης που προστατεύονται και που είναι περιφερειακής, ε, τοπικής μάλλον ε, ε, παραγωγής οι μικρομεσαίε μα επιχειρήσει προστατεύονται, οι γεωργοί μα προστατεύονται, οι συμπολίτε μα προστατεύονται. Ε, αυτό είναι το ερώτημα. Πού βρισκόμαστε σήμερα, πού θα μπορούσαμε να είμαστε αύριο με τη ΣΕΤΑ. Ίσως η ΣΕΤΑ να μπορεί να τελειοποιηθεί και μάλιστα υπάρχουν διάφορες ρήτρε όπω η ρήτρα ασφαλεία ή ο κατάλογο τη αναθεώρησης για κάποιε ονομασίε. ναι, μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να προστατεύσουμε, αλλά η ΣΕΤΑ ε, επιδεινώνει την κατάσταση, τη βελτιώνει. Τη βελτιώνει Κάθε μέρα που χάνουμε λοιπόν πριν να απογραφεί αυτή η συμφωνία είναι μια μέρα χαμένη για τις επιχειρήσεις μας, για τους γεωργού μας και για τους συμπολίτε μας. Ελπίζω πραγματικά πως θα επιταχυνθεί το χρονοδιάγραμμα και ότι θα μπορέσουμε νυφάλια αφού θα έχουμε λάβει τις απαντήσεις ίσως αλλάζοντας το περιθώριο για το ΙΣΕΣ e με την προσωρινή εφαρμογή. Όχι, δεν ισχύει και σύμφωνα με τον κύριο Μανιέτ υπάρχει και μια προθεσμία για τον ορισμό των δικαστών. Μπορούμε να δουλεύουμε δουλέψουμε ναι, για την βελτίωση του κειμένου, αλλά οι 1500 σελίδες είναι μια ε, συμφωνία που κερδοφόρο για την Ευρώπη και κερδοφόρο για τον Καναδά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτή η συζήτηση για τις εμπορικές συμφωνίες δεν είναι μόνο για να πούμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε εμπορική πολιτική. Είναι για να δείξουμε κιόλας ότι είναι παραδοσιακή πολιτική αυτή των εμπορικών συναλλαγών για να μειώνονται οι δασμοί και τα άλλα εμπόδια και επεκτείνεται τώρα σε διάφορους τομείς που απαιτούν το δημοκρατικό έλεγχο. Είναι λάθος να επενήσεται κανείς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι δημοκρατικό όργανο αυτό που είπατε και εσείς το υπογραμμίζω. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει και να αναλάβουμε τις ευθύνες των καθηκόντων που έχουμε. Και με δυσφορία βλέπω ότι πολλές φορές ε, ζητήματα τα οποία έπρεπε να μας απασχολήσουν εδώ στο Κοινοβούλιο ε, και να δοθούν απαντήσεις από τα κράτη-μέλη δεν ε, λύθηκαν πριν ε, από τι 12 παρα 5 ουσιαστικά, πριν ακριβώ από την υπογραφή τη συμφωνία και έτσι δεν δόθηκε ποτέ, ποτέ ουσιαστική ευκαιρία για συζήτηση εδώ. Και βεβαίω θέλω να δοθούν διευκρινήσει, έχουν απόλυτα κρίσιμη σημασία. Να γνωρίζει ο κόσμο τι ψηφίζουμε. Αυτό που βλέπω με δυσφορία επίση είναι ότι οι λεγόμενε διευκρινήσει μάλλον περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Φιλιππίν, δηλώσεις της Σλοβενίας, Πολωνίας και Βελγίου που ζητούν τώρα αλλαγές στο κείμενο της συνθήκης για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ επενδυτών κρατών ή το σύστημα αυτό των διαιτητικών δικαστηρίων. Και η Επιτροπή λένε όχι δεν ξανανοίγουμε το κείμενο. Τι ψηφίζουμε ακριβώς τότε γιατί το Βέλγιο ήταν απόλυτα σαφές και άλλα κράτη επίσης δήλωσαν ότι αν δεν τηρηθούν οι διακηρύξεις θα ασκήσουν το δικαίωμα της αρνησικυρίας. Πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις σχετικά με το σύστημα της διαιτησίας πριν φτάσουμε στην ώρα των ψηφοφοριών στα Εθνικά Κοινοβούλια για την κύρωση και τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Διεθνικής διευθέτηση των Διαφορών. Και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι θα πούμε εάν μετά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο βρεθούμε εκτεθειμένοι και δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε αυτά τα οποία έχουμε διακήρυξει. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς λοιπόν ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε, πώς εμπλέκεται το Κοινοβούλιο και τι συμβαίνει εάν όταν προχωρήσουμε και έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία δεν έχουν ακόμη δοθεί οι κατάλληλες απαντήσεις στα μελήματα που εκφράζονται. Επίσης, η Σύμβαση της Βιέννης που τακτικά επανέρχεται, κάνει μια σαφέστατη ιεράρχηση μεταξύ των διαφόρων ειδών διεθνών συμφωνιών. Μεταξύ αυτών λοιπόν των διακήρυξεων, ερμηνευτικών δηλώσεων, πρωτοκόλων και όλα αυτά, υπάρχει μια ιεράρχηση σε σχέση με το κείμενο της συμφωνίας και συμφωνώ με τη Σκάκελερ ότι χρειάζεται σαφής ανάλυση από πλευρά της Επιτροπής. Τι είναι νομικά δεσμευτικό, τι συνέπειες έχει το κάθε και θα φτάνω στην τρίτη παρατήρηση, ότι διαπιστώνω αντιφάσεις φερρυπίν μεταξύ διαφόρων δηλώσεων και ερμηνευτικού, του ερμηνευτικού μέσου, του ερμηνευτικού πρωτοκόλου που λέει ότι θα υπάρξει έγκριση των αποφάσεων από την Μεκτή Επιτροπή ε, ΣΕΤΑ, η οποία θα λάβει τις σχετικές ερμηνευτικές ε, διατάξεις. Αυτό είναι που με ανησυχεί περισσότερο ακόμη σε σχέση με το ερμηνευτικό. Δηλαδή τα εργασιακά δικαιώματα, οι διαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας καθίστανται έτσι δεσμευτικές. Θα έχουμε ένα κεφάλαιο πραγματικής ανάπτυξης και αηφορίας. Και τέλει, η συμφωνία που κυκλοφόρησε και νομίζω η δήλωση σε σχέση με, τη συνταγματική, με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας που λέει η Επιτροπή δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια απόφαση στο μέλλον. Εδώ έχουμε μια ε, ευθεία αντίφαση μεταξύ δύο κειμένων διεθνούς συμφωνίας ή διεθνού, διεθνούς νομοθετήματος. Μέχρι να ξεκαθαριστεί αυτή η ιεραρχική σχέση μεταξύ των δύο κειμένων, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε τι συνέπειε έχει το καθετή και για μένα αυτό δεν συνιστά σωστή ε, ρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Όμπερμαϊερ. Ναι, ήδη επισημάνθηκε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι συνάδελφοι κουράζονται από την επαναληπτική κιόλας αλλά πρέπει να δούμε πλέον τα αποτελέσματα. Πρέπει να δούμε αποτελέσματα που θα γίνονται και αποδεκτά, θα γίνουν και αποδεκτά σε επίπεδο κοινοβουλίου για να εγγραφούν στην, ε, στην ε, συνθήκη. Γιατί κατά τα άλλα μόνο εργασιοθεραπεία κάνουμε. Πρόκειται λοιπόν να προχωρήσουμε και σε ψηφοφορίε στα κράτη-μέλη. Πρέπει να γνωρίζουμε τι κάνουμε, πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και σε ποιο βαθμό τα έχουμε επιλύσει. Και αυτό θα είναι για μένα κρίσιμο και για του βουλευτέ μα, βέβαια, στην Αυστρία, αγαπητοί συνάδελφοι, για να εγκρίνουν. Άρα είναι καλό να εγείρονται τα ζητήματα. Δεύτερον, ενδιαφέρον το ότι Κάποιοι ζητούν συγγνώμη επειδή έχουν κάποιες επιφυλάξεις ε, ή ανησυχίες. Αχ, με συγχωρείτε, δεν ήθελα να είμαι τόσο λαϊκιστή. Μα με συγχωρείτε, εμεί οι βουλευτέ είμαστε υποχρεωμένοι να διατυπώνουμε ερωτήσει, να έχουμε μελήματα και ανησυχίε και να εκπροσωπούμε έτσι τα μελήματα και τι ανησυχίε των πολιτών. Και πρέπει να συγχαρούμε του βαλόνου που είχαν το θάρρο επί τη βάση των συνταγματικών του δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων να εγείρουν τα ζητήματα αυτά και να καθυστερήσουν τη διαδικασία. Γιατί νομίζω ότι έτσι εκφράζουν τα μελήματα και τις ανησυχίες ε, που και στην Αυστρία θα έπρεπε να έχουν εγερθεί. Και επίσης κάποια ζητήματα τα οποία δυστυχώς δεν καλύπτονται και αφορούν όλο αυτό το πλέγμα ε, τις βασικές αρχές δηλαδή που ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρουν και τους πολίτες μας που είναι αρχές της Ευρώπης, η αρχή της πρόληψης πάνω απ' όλα που ναι, κάποιοι συνάδελφοι λένε Α, κοιτάξτε, είναι προδιαγραφέ αυτέ δικέ μα που τόσο ή πρέπει να τηρηθούν, δεν τίθεται ένα αμφιβόλο κτλ. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά θα ήταν πολύ καλύτερο να είναι σαφώς διατυπωμένη μέσα στο κείμενο ως θεμελιώδης αρχή αυτή η αρχή της πρόληψης. Επίσης, η κανονιστική, η ρυθμιστική αρχή, regulatory principle, που έχει μεγάλη σημασία. Το τέτοια που ίσως δεν μπορούμε ακόμα καν να την εκτιμήσουμε στο σύνολό της. Εδώ βλέπουμε να κινείται ένα φάσμα φόβου και απειλής, χωρίς όμως μια πραγματική εκτίμηση των συνεπειών. Καλό θα ήταν να συζητούμε για το, πραγματικά, για το πραγματικό αντικείμενο των ρυθμίσεων και όχι για το τι νομίζουμε ότι μπορεί να ρυθμίζεται. Όλα αυτά λοιπόν που κάποιοι ονομάζουν λαϊκιστικές ε, ε, φωνές ε, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά πραγματικά και γνήσια μελήματα στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριο Σφιέναρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πραγματική ουσία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συγκεντρώνει την κυριαρχία. Και αυτά τα έχουμε συζητήσει. Για παράδειγμα, σε θέματα μετανάστευσης, άμυνα και ούτω καθεξής. Πολλά από αυτά που συζητούμε τώρα. Κάποιοι έξυπνοι κάθισαν όμως, κάποιοι φύσοι άνθρωποι δηλαδή, κάθισαν το 1957 και σκέφτηκαν ότι ίσως μια ε, τελωνιακή ένωση να ήταν καλή και εκεί θα χρειαζόταν να συγκεντρωθεί κυριαρχία σε ένα, σε ένα συγκεντρωτικό επίπεδο και μετά προέκυψε ευημερία. Μέχρι τώρα όμως. Διότι τώρα πολλοί αρχίζουν και διαρωτώνται αν δεν θα πρέπει να ξαναπάρουν πίσω την κυριαρχία από το ευρωπαϊκό επίπεδο και να τα επανεθνικοποιήσουν και να ψηφίζουν όχι μόνο οι εθνικές βουλές αλλά και οι περιφέρειες των χωρών τους. Αυτό όμως θα είναι καταστροφικό και για την εμπορική πολιτική και για την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρά εκεί όπου έχει καταρχήν αρμοδιότητα. Όταν η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική βρίσκεται σε αυτά τα χάλια, νομίζω ότι είναι και νομιμοποιείται να θέσει κανεί την ερώτηση αυτή. Αν ακολουθήσουμε δηλαδή αυτόν τον δρόμο, τότε θα πούμε ότι και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει την ε, δημοκρατική νομοποίηση. Ε, εγώ άκουσα και τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Μάλμστρομ. Είπε ότι υπάρχουν ορισμένες νομικές αβεβαιότητες σχετικά με την αρμοδιότητα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είναι υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συνθήκη αυτή, ε, συμφωνία δηλαδή. Εμείς ωστόσο εδώ οι ευρωβουλευτές διαβάζουμε τις συνθήκες και θεωρούμε ότι εμείς έχουμε την αρμοδιότητα να το κάνουμε. Όμως για πολιτικούς λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν τη σοφία της, το βάζω αυτό εισαγωγικά, αποφάσισε ότι είναι μεικτή, μεικτή η αρμοδιότητα. Ορισμένοι το κράβγασαν και είπαν ότι ήταν καλή η απόφαση αυτή. Αυτοί όμως αμφισβητούν τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι νόημα έχει να γίνονται όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις όπου και εγώ έχω πάει 12 χρόνια τώρα εάν η πολιτική σε αυτή απόφαση είναι καλή. Ακούω ακόμα και τα έχω ακούσει πολλές φορές. Λένε, α, θέτουμε απλώς ερωτήσεις. Μπράβο, καλά κάνετε, λέω εγώ. Οι πολίτες θέτουν ερωτήσεις. Εγώ μεταφέρω τις ερωτήσεις των πολιτών εδώ. Να κάνω και μια προσθήκη στρατηγική αυτή. Πώς θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις αυτές. Τι θα λέγατε να συναντούμε τους πολίτες και να τους εξηγούμε. Δεν ξέρω πόσες εμπειρευμένες δηλώσεις έχουν ε, εκδοθεί ήδη. Θα έλεγα εγώ ότι πρόκειται για αυτό το SETA for Dummies. Είναι βέβαια περίπλοκο το κείμενο του SETA, όμως υπάρχουν τόσες ερμηνευτικές δηλώσεις για χίλια δύο θέματα που άπτονται της συμφωνίας. Όμως και πάλι ακόμα εδώ και στην παρούσα αίθουσα τίθεται ξανά και ξανά οι ίδιες ερωτήσεις. Γιατί δεν διαβάζετε το κείμενο της ΣΕΤΑ, τις ερμηνευτικές δηλώσεις, αντί και έτσι να απαντήσετε ερωτήσεις, αντί να τις επαναλαμβάνετε τις ερωτήσεις. Αυτοί που επαναλαμβάνουν τις ίδιες και τις ίδιες, ε, τους ίδιους και τους ίδιους εσφαλμένους χειρισμούς για τις δημόσιες προβλήσεις τα Και, και θέτουν ερωτήσεις. Μα γιατί δεν βρίσκουν τις απαντήσεις που είναι μέσα στο κείμενο. Τώρα, το θέμα της προστασίας των επενδύσεων. Ακούσαμε πάλι σήμερα εδώ κάποιους να λένε ότι ανησυχούμε για πρώτη φορά που δίνουμε τη δυνατότητα της ιδιωτικής δικαιοσύνης και οι Βαλόνοι αντελήφθησαν επιτέλους τώρα ότι υπάρχει κάτι που λέγεται προστασία επενδύσεων και μας ανησυχεί. Μα πρόκειται για καλαμπούρι. Το Βέλγιο έχει 60, 60 διμερείς συμφωνίες που περιλαμβάνουν και συστήματα και συστήματα διαιτητικής επίλυσης διαφορών γιατί ενισχύουν τόσο πολύ. Μια φορά έγινε προσφυγή εναντίον τους και κέρδισαν. Έχουν δύο νέες διμερείς συμφωνίες από το 2009, Παναμά και Τατζικιστάν. Γιατί δεν ξεσηκώθηκαν οι βαλόνοι κατά αυτών των συμφωνιών, γιατί δεν έγινε συζήτηση. Ακούσατε ποτέ να λένε ότι θέλουμε να διαγράψουμε όλες τις παλιές συμφωνίες, όχι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ίσως θα πρέπει να ρωτήσω την κυρία Αρενά που ήταν και υπουργό στη βελική κυβέρνηση όταν συμφώνησαν με το Τατζικιστάν και τον Παναμά με κεφάλαια για διαιτητική επίλυση διαφορών με τη βελική κυβέρνηση. Τι πρόβλημα υπάρχει εκεί. Γιατί ξεπήδησε τούτο το πρόβλημα εδώ, σε αυτή τη συνθήκη μόνο και την τελευταία στιγμή. Εγώ νομίζω ότι και το Βέλγιο το ίδιο είχε πλήθος ευκαιριών να βρει τις απαντήσεις τη ερωτήσεις. Ενδιαφέρομαι να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσες φορές η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε για την ΣΕΤΑ στο Συμβούλιο και πόσες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πόσες φορές έχετε απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερωτήσεις. Διότι ίσως τελικά να μην έχει και διαφορά είτε έλθετε είτε όχι, διότι προφανώς ο κόσμος δεν σας ακούει. Λούνς. Ευχαριστώ. Είμαι και εγώ Βέλγος Ευρωβουλευτής, αν και δεν είμαι βαλόνος είμαι Φλαμανδός. Η Φλάνδρα δε είναι υπέρ της ΣΕΤΑ. Το δε κόμμα μου, το ΕΝΒΑ, το μεγαλύτερο κόμμα στη Φλάνδρα και στην Βελγική και στο Βέλγιο γενικότερα, διακόπτει η κυρία Αρένα. Πρέπει να απαντήσω και αλλιώ ε, θα μιλήσετε και άλλα πράγματα εκτός από το Βέλγιο μόνο. Βρίσκω εντάξει, κάποια φάση θα μου δώσετε δυνατότητα να απαντήσω. Εντάξει, να κάνουμε συζήτηση για το Βέλγιο, άμα θέλετε. Ήσυχα, ήσυχα. Έχει ο καθένα το δικαίωμα να λάβει το λόγο. Ο κύριο έχει το λόγο. Εφόσον θα ήθελε να περιμένει η κυρία Αρενά, θα αντιληφθεί ότι δεν πρόκειται για επίθεση εκ μέρου μου, αλλά για ενθάρρυνση. Είπα ότι είμαι και εγώ Βέλγο Ευρωβουλευτή και λαμβάνω το λόγο για λογαριασμό ενό σημαντικού βελγικού κόμματο. Η Βαλονία λοιπόν έχει κάθε δικαίωμα να πράξει αυτό που έπραξε. Κάθε δικαίωμα θεωρώ εγώ. Η Βαλονία είναι δημοκρατικό φόρουμ, άλλωστε και αρκετά μεγάλο θα έλεγα εγώ και νομίζω ότι πάντοτε συμφωνούσαμε άλλωστε σε αυτό ότι χρειαζόμαστε περισσότερη δημοκρατία. Και αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα άσκησε η Βαλονία. Έχει δικαίωμα να το πράξει αυτό. Και χαίρομαι άλλωστε που βλέπω ότι συμφωνεί και η πολιτική της ομάδα. Ότι δηλαδή οι χώρες μέλη έχουν σημαντικό ρόλο στην συζήτηση αυτή. Δεύτερο, αυτό που είδαμε τώρα στην πιο πρόσφατη συζήτηση που ήταν της τελευταίας στιγμής, πρόσφερε ωστόσο ένα πλεονέκτημα, δηλαδή ότι η επικοινωνία μας σήμερα διευκολύνεται. Ο κύριος Φιέλνερ σωστά είπε ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που κυκλοφορούν, λίγες όμως απαντήσεις. Και νομίζω ότι σήμερα προστίθεται ένα ακόμη επιχείρημα, δηλαδή η επικοινωνία που προήλθε από τη βαλονική στάση. Και η ανακοίνωση της Βαλωνίας δίνει κάποιες απαντήσεις. Μας παρομοιάζουν ορισμένοι με το μικρό εκείνο γαλατικό χωριό, εδώ, τη Βαλωνία δηλαδή. Όμως την ανακοίνωσή τους λένε ότι η συμφωνία ΣΕΤΑ δεν θα οδηγήσει στο να καταναλώνουμε κρέας με ορμόνες. Λένε επίσης ότι το κοινωνικό μας μοντέλο παραμένει ισχυρό. Λέει επίσης η ίδια ανακοίνωση ότι οι κοινωνικές μας υπηρεσίες προστατεύονται. Δεν τα λέω εγώ αυτά, ούτε η ΣΕΤΑ, τα λέει η ίδια η Βαλονία στην ανακοίνωσή της. Λέει επίσης ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ιδιωτική δικαιοσύνη. Δεν το λέω πάλι εγώ, το λέει η Βαλονία στην ανακοίνωσή της. Πέμπτο, λέει ότι ούτε ανοίγεται η πόρτα σε δούριο ύπο των ε, πολυεθνικών. Τα λέει αυτά η ανακοίνωση της Βανωνίας, του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Έκτο, λέει ότι προστατεύονται τα εθνικά προϊόντα. Έβδομο, οι τοπικές γεωρικές παραγωγές, τα διατροφικά μας προϊόντα. Πάλι η Βαλονία τα λέει αυτά. Όγδο, διευκολύνονται οι εξαγωγικές δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία απασχολούν στη συζήτηση αυτή και τώρα όλα αυτά διευκολύνονται. Διότι ακριβώς οι βαλόνοι ξεσηκώθηκαν, αντιστάθηκαν και καταλήξαμε σε αυτή την ανακοίνωση. Και μάλιστα όλα αυτά χωρίς να έχει αλλάξει ούτε ένα γράμμα στο κείμενο της ΣΕΤΑ. Μου φαίνεται λοιπόν ότι δίνονται απαντήσεις. Θέσανε ερωτήσεις έλαβαν απαντήσει και δίνουν απαντήσει. Δεν θα υπάρξει νέα σέτα. Και στα αγγλικά να σα το πω. There is no new SETA. Δεν έχει ανάξει ούτε ένα γράμμα στο κείμενο της συμφωνίας. Συζητείται το ISDS ή ICS, τέλο πάντων το σύστημα διευθυντική επίλυσης των διαφορών επενδυτών και κρατών. Επιβάλλονται κάποιοι όροι, ναι, έχει καλώς, αλλά στην ουσία πρόκειται για μια ενίσχυση των όσων γνωρίζουμε ήδη ότι δεν θα υπάρξει ιδιωτική δικαιοσύνη. Ναι, θα είναι ανεξάρτητοι δικαστές. Αλλά είναι κάτι το οποίο συζητούμε εδώ και καιρό και μήνες. Δεν είναι λοιπόν νέα συζήτηση αυτή. Τα γνωρίζουμε αυτά όλα. Αλλά τα διαλαμβάνει εκ νέου, ρητά, η βαλονική ανακοίνωση. Και γνωρίζουμε επίσης περί τίνος πρόκειται και γνωρίζουμε και τι θα ψηφίσουμε. Είναι πράγματα που γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Και τέλος, μόλις κατέβηκα από το αεροπλάνο, επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου παρακολούθησα τις Αμερικανικές εκλογές, άκουσα και τον πρώτο λόγο του νέου Προέδρου και μπορώ να φανταστώ ότι η αριστερή, η άκρο αριστερή και οι πράσινοι θα είναι χαρούμενοι από το αποτέλεσμα, διότι δεν είναι πλέον μόνοι τους στον αγώνα κατά του ελεύθερου εμπορίου και υπέρ του προστατευτισμού και απομονωτισμού. Επιτέλους βρήκαν κάποιον που θα του συμπαρασταθεί, τον κύριο Τραμπ. Ακούγοντας τον, την πρώτη ομιλία στην Νέα Υόρκη του Τραμπ, βεβαίως μου φάνηκε πολύ πιο μετριοπαθής. Θα δούμε τώρα εάν η καυτή σούπα που έφτιαξε στην προεκλογική θα καταναλωθεί το ίδιο καυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτς τελευταίος, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Βαθύτατη ανησυχία αισθάνομαι μετά τα τελευταία μάλιστα λόγια για να ξεκινήσω με αυτό σε σχέση με αυτόν τον νέο πρόεδρο. Και με τη σύγκριση που ακούσα από τον κύριο Λούνες. Ακριβώς αυτό είμαστε στο κέντρο, στο επικέντρο της συζήτησης. Πολιτικές θέσεις για το πώς θα λειτουργήσει η ΣΕΤΑ σε κοινωνικό επίπεδο, αν θα είναι πιο ε, ανοιχτή, ε, αν θα καλυφθούν ε, τα διάφορα μελήματα. Βεβαίως είναι και αυτό ένα ζήτημα και με τη νέα αυτή συμφωνία τελικά έχουμε να κάνουμε με τον τρόπο της οργάνωσης της λειτουργίας των οικονομιών μας. Με τεράστιες και κοινωνικές βέβαια συνέπειες. Και αυτό ακριβώς είναι ο λόγος της συζήτηση και στα κράτη-μέλη και στον Καναδά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση δημόσιο διάλογο στον Καναδά, μην το ξεχνάμε. Και εμεί τώρα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινούμε με ένα κείμενο που έχει συμφωνηθεί, που έχει υπογραφεί, να ασχολούμαστε με βάση την νομοθεσία ενώ έχουμε πιο νωρίς ακόμη αρχίσει και ζητήσει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, διεκδικώντας ένα δημοκρατικό δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακριβώς επειδή θέλουμε να φέρουμε τη φωνή μας τη δημοκρατική σε αυτές τις πολιτικές και νομικές εξελίξεις. Για να μην αφήσουμε εθνικιστικά ή περιφερειακά συμφέροντα να απορδιαρθρώνουν μια συμφωνία που μπορεί να είναι για το καλό όλων, αλλά να έχει τη δυνατότητα ο κόσμο μέσα στι χώρε και τι περιφέρειες να συμμετάσχει στην, στο πολιτικό γίγνεσθε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ζητούμενο και ισχύει και για τη ΣΕΤ όπω και για κάθε άλλη διεθνή εμπορική συμφωνία με πολλέ διαφορετικέ πολιτικές τοποθετήσεις, αντιφάσεις και διαφωνίες και είναι σωστό, είναι λογικό, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν οι αμφιβολίες και οι αντιδράσεις. Πρέπει να μπουν στη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει να κάνει άλλωστε και με το χαρακτηρισμό μιας συμφωνίας ως μεικτή σημή. Είπε το Σταγματικό Δικαστήριο, τουλάχιστον για μας, τη γερμανική σκοπιά δηλαδή, ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι μόνο από πλευράς μόνο σε γερμανικό επίπεδο μπορούν να αποφασιστούν, μόνο από τη Γερμανία δηλαδή, όπως η εισαγωγή των διαιτητικών αυτών δικαστηρίων για την επίλυση των διαφορών. Το ερωτηματικό όμως που γεννάται τώρα για μας ως Ευρωπαίους πολιτικούς και για την ευρωπαϊκή πολιτική έχει τεράστιες συνέπειες ως προς τη λειτουργία της ΕΤΑ ως συμφωνίας στο μέλλον. Και αυτό πρέπει να επαληθεύσουμε και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση, το ότι ακούμε κάποιες απαντήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν και νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις επιλογές Επιτροπής στο τελευταίο διάστημα. Και για να γυρίσω στη συζήτηση και να τοποθετηθώ σε αυτά που αν και ο Ντάνελ και ο Κρίστοφερ να υπάρχουν πολλά σημεία ή θεωρήσεις που μπορεί να είναι επικριτικές, διαφορετικές θέσεις που δεν έχουν συγκεραστεί. Εμείς, σε παραδείγματι, εμείς βλέπουμε επικριτικά το, την προσέγγιση ενός αρνητικού καταλόγου από τη δική μας την πολιτική τοποθέτηση. Γι' αυτό το γύρουμε ως θέμα στη συζήτηση, γιατί βλέπουμε ένα κίνδυνο σε σχέση με την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, Φερρυπή. Εμείς, παραδείγματι, τασόμεθα υπέρ της αρχής της πρόληψης. Τώρα έχουμε μια συμφωνία με συνέπειες έναντι των οποίων πρέπει να βγούμε στην κοινωνία, να τις συζητήσουμε και να πούμε τι, τι, σημαίνουν. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Και τρίτον, για την εσωτερική συζήτηση σχετική με το Βέλγιο. Μα είναι πονδιακό κράτος το Βέλγιο. και συζητήθηκε το ζήτημα με σοβαρότητα. Ο κάθε υπουργό, πιστεύω, θα έπρεπε στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου και των αρμοδιοτήτων του να είναι βέβαιο ότι κάθε τομέα έχει καλυφθεί ικανοποιητικά και να γίνει βεβαίω στη συνέχεια και μετά η διαβάθμιση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι κομμάτι, ποιο κομμάτι ανήκει στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, αλλά ταυτόχρονα και κάθε αποφάση που θα, γίνει σε τοπικό, θα ληφθεί σε τοπικό ή άλλο επίπεδο, σε ποιο βαθμό επηρεάζει το ευρωπαϊκό ή μη. Αυτό πρέπει να συστήσουμε, αυτό πρέπει να προβάλλουμε. Αυτή είναι η ενδυνάμωση συζητησουμε αυτο πρεπει να πολίτη, η δυνατότητα δηλαδή για τον πολίτη να μπει στο δημοκρατικό γίγνεσθε για να γίνει ο πραγματικός διάλογος και να μην τον παραδώσουμε στα χέρια μόνο των λαϊκιστικών δυνάμεων. Χρειάζεται η παρακολούθηση αυτή, η δημοκρατική των εξελίξεων. Και γι' αυτό θα ήθελα για όλους αυτούς που μιλούν για δημοκρατία και λοιπά Να πω ξεκάθαρα ότι είναι καθήκον μας και πρέπει με σοβαρότητα να το επιτελέσουμε. Μακάρι να είχαμε τη την, ε, να την ευκαιρία, να είχαμε το θάρρος να συστήσουμε την υπόθεση αυτή και σε άλλους χώρους με σοβαρότητα. Και πιστεύω, ελπίζω τουλάχιστον ε, το ψήφισμα να καταγράψει ένα ευρύ φάσμα θέσεων από πλευράς των ομάδων και να αποτελέσει ένα καλό συνοδευτικό έγραφο τη συμφωνία ΣΕΤΑ και της κύρωσης τουλάχιστον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ η Καρολίν για να τελειώνουμε. Ναι, ευχαριστώ. Δυστυχώς με λησμονήσατε. Στη συζήτηση αυτή λοιπόν, στη συζητήσει όλε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, δυστυχώς λησμονούμε ότι υπάρχουν διαφορετικέ πραγματικότητε, πολλά ερωτηματικά στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις προκειμένου να ληφθούν και οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει ως εκ τούτου να αναλογιστούμε γιατί γεννήθηκαν όλα αυτά τα ερωτηματικά, γιατί ήταν τόσες ασάφειες. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχαμε τη δυνατότητα της παρέμβασης στις ε, διαπραγματεύσεις. Δεν αρκεί ένα ψήφισμα για να ληφθεί υπόψη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής η δική μας θέση. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να πούμε ναι ή όχι. Ναι μας κάνει, ναι ε, δεν μας ικανοποιεί. Δεν έχουμε την ευκαιρία και το χρόνο να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες και να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες συμφωνίας. Αυτό θα έπρεπε να έχει συμβεί. Απαριθμήθηκαν ε, τώρα τα ζητήματα, επί παραδείγματι το θέμα του, ε, του διαιτητικού συστήματος επίλυσης των διαφορών και όλων των ε, ερμηνευτικών και άλλων δηλώσεων που προσαρτώνται στη συμφωνία που δεν δίνουν όμως ακριβείς απαντήσεις. Και μετά την απόφαση για τον Brexit παραμένουν πολλές εκκρεμότητες άλλες, πάλι στις οποίες θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να εξετάσουμε πώς θα προχωρήσουν, τι εξέλιξη και τι συνέπειες θα δώσουν. Επίσης μην ξεχνάμε ότι έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολεί τους πάντες, έχουν ενημερωθεί. Χρειάζεται ίσως ε, ε, να ξεπεράσουμε το στάδιο του να εξηγήσουμε τι σημαίνει ΣΕΤΑ, αλλά να δούμε την ουσία της υπόθεση και τον τρόπο με τον οποίο θα ταχθούμε τελικά ως Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Μαώρο. Απαντήσεις χρειάζονται, όπως βλέπετε. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, να ζητήσω συγγνώμη που άργησα. Έρχομαι από, προέρχομαι από μια πόλη χαλιβουργική και μεγάλωσα στην Ιταλία τη δεκαετία του 60 και 70 και γι' αυτό και σέβομαι πολύ τους χαλιβουργούς ε, με, με εντυπωσίασε που είδα τέσσερις ηλικιωμένου πολίτες να διαδηλώνουν έξω από το <laughs> κτίριό μου και να μου λένε ότι δεν μπορώ να βγω γιατί ε, διαδήλωναν λέει αυτοί οι τέσσερις ηλικιωμένοι και δεν ήταν ασφαλές για μένα. Τέλος πάντων, πολύ προστασία. Τώρα, συνοψίσατε κάπω τα πράγματα. Εγώ θα προσπαθήσω να σα δώσω όσο γίνεται περισσότερο αντικειμενικά τα στοιχεία. Εάν μου, αν ξεχάσω κάτι, δεδομένων των χρονικών ορίων, είμαστε σε επαφή με πολλού ε, από τα μέλη τη Επιτροπή και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό ευχαρίστω, να σα δώσω και άλλε διευκρινήσει. Ρωτήθηκε, ε, θέθη ερώτηση για το πώς έγιναν αυτές οι δηλώσεις. Η Κομισιόν δεν έκανε τίποτα παράξενο ή καινούριο ως προς αυτό το στοιχείο. Ήταν ίσως πιο δραματική η κατάσταση από ό,τι ήθεστε. Αλλά έχουμε ρόλο διευκόλυνσης της διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα κράτη-μέλη και πάμε όταν μας το ζητούν. Έχουμε, ας πούμε, χρειάστηκε να συζητήσουμε μετά από αίτημα της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης να συζητήσουμε για θέματα όχι μόνο με τους υπουργούς αλλά και με τους υπουργούς των διαφόρων κρατηδίων που το επιθυμούσαν. Ε, τις τελευταίες εβδομάδες της συζήτησης περί ΣΕΤΑ ήμασταν σε στενή επαφή με τουλάχιστον μισ, ε, μισή ντουζίνα κράτη-μέλη που έχουν περάσει την συμφωνία από τις εθνικές κυβερνήσεις. Μόνο στην περίπτωση του Βελγίου μας ζητήθηκε να ε, έρθουμε σε επαφή με την περιφερειακή κυβέρνηση. Το κάναμε αυτό κατόπιν αιτήματος της Βελγικής Ομοσπονδικής Κυβέρνησης. Ξέραμε ότι η βαλλονική κυβέρνηση ήταν υπέρ και ήταν πολύ παραγωγική ε, δουλειά. Ο ρόλος της Κομισιόν είναι να εξηγεί, να διευκολύνει και οποτεδήποτε οι εξηγήσει μας δεν αρκούσαν, προσπαθήσαμε να προσθέσουμε είτε μαζί με τους Καναδούς μέσω του κοινού ερμηνευτικού μέσου, είτε μέσω των ευρωπαϊκών δηλώσεων και με αυτό σε αυτό περιλαμβάνω δηλώσεις της Κομισιόν, δηλώσεις του Συμβουλίου, κάποιες από τις δηλώσεις μεμονωμένων κρατών μελών, αλλά θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Τώρα, για την φύση αυτού του μέσου, όπως ορισμένοι από την Επιτροπή είπαν, κάποιοι βουλευτές είπαν, Αυτά ε, είναι ερμηνευτικό μέσο. Η νομική αξία του ορίζεται στη δήλωση Παριθμού 38 που έχει γίνει από τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Με αυτήν την δήλωση συμφωνούμε. Εμείς συνυπογράφουμε αυτήν τη δήλωση νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Δεν είναι αλλαγή στη ΣΕΤΑ, αλλά είναι διευκρίνηση. Και είναι μια διευκρίνηση που, όπως λέει, η νομική υπηρεσία έχει νομική ισχύ. Είναι μια ερμηνευτική δήλωση με νομική ισχύ. Όποιος θέλει να ερμηνεύσει την ΣΕΤΑ, εάν δεν την βρίσκει σαφή, θα δεσμεύεται από τις δηλώσεις που έχουν εκδώσει τα μέρη ως την αυθεντική ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων κάθε φορά. Έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε και ένα πίνακα συμφωνίας. Ε, δεν είναι πλήρης, αλλά είναι αρκετά περιστατωμένος για να δούμε ε, με παραπομπές ε, το κείμενο της συμφωνίας. Αυτό έγινε κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματο της κυβέρνησης της Βαλωνίας για τα σημεία που επικρατούσε αβεβαιότητα. Τώρα, οι ευρωπαϊκές δηλώσεις ε, επίσης σύμφωνα με την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου αποτελούν κομμάτι του ερμηνευτικού συμπλέγματος. Είναι μονομερείς για κάποιον Ευρωπαίο φορέα, αλλά αφορούν θέματα τα οποία δεν έχουν ε, νόημα γιατί ο Καναδά, ας πούμε, πρόληψη προφύλαξη μάλλον. Η προφύλαξη αναφέρεται μέσω σε μια ερμηνευτική δήλωση Δηλαδή, ο Καναδάς και η Ένωση επιβεβαιώνουν την αρχή της προφύλαξης όπως εκφράζεται στις διεθνείς συμφωνίες που τα δύο μέρη έχουν υπογράψει. Σε μια διεθνή συμφωνία, εάν ένα θέμα δεν αναφέρεται, αυτό σημαίνει πως ισχύει η απαράλλακτη εγχώρια νομοθεσία του μερών. Για να είναι αυτό απόλυτα σαφέ, κάναμε και μια δήλωση που εξηγεί ότι τίποτα στη ΣΕΤΑ δεν παρεμβαίνει ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί αρχής της προφύλαξης και όπως όλοι γνωρίζουμε αυτή η αρχή της προφύλαξης είναι γεγραμμένη στις συνθήκες και είναι καθήκον κάθε ευρωπαϊκού θεσμού και των, των κρατών μελών να την εφαρμόσουν. Τίποτα στη ΣΕΤΑ δεν μας εμποδίζει να το κάνουμε αυτό. Γιατί δεν υποχρεώνουμε τον Καναδά να δεχτεί μια αρχή την οποία δεν έχουν εκεί θεσπισμένη, όπως και εκείνος δεν μας δέχτηκε να την αναιρέσουμε. Δηλαδή ο σεβασμός στις αρχές είναι αμοιβαίος. Παρόμοια ερμηνευτική αξία των δηλώσεων έχουμε λοιπόν σε σχέση με τους διάφορους φορείς. Το κοινό μέσο είναι, υπάρχει για να δεσμεύσει τον Καναδά σε αυτή την ερμηνεία. Οι δηλώσεις από τους Ευρωπαίους ε, εταίρους ε, δεσμεύουν τους ίδιους σε θέματα που αφορούν όχι τον Καναδά, αλλά το πώς οι Ευρωπαίοι ε, φορείς θα εφαρμόσουν την συμφωνία. Υπάρχει ένα στοιχείο αμφισημίας και όπου γίνονται οι μονομερείς δηλώσεις από τα κράτη-μέλη. Εκείνες είναι δηλώσεις των κρατών μελών Ορισμένες από αυτές έχουν, με την επιλογή των ε, ενδιαφερομένων κρατών έχουν συζητηθεί με την Κομισιόν και το Γραμματεία του Συμβουλίου. Άλλες έχουν εκδοθεί υπό την απόλυτη ευθύνη των ε, λόγω κρατών μελών. Για αυτές δεν μπορούμε να σχολιάσουμε ούτε για την ακρίβειά τους, ούτε για το στόχο τους. Δεν ήμασταν μέσα στη συζήτηση, δεν συμμετείχαμε καν στη συζήτηση. Όταν μας συμβουλέθηκαν τα κρατημέλη, εμείς ε, ε, τους συμβουλέψαμε έτσι ώστε ό,τι και αν δήλωναν τα κρατημέλη να ταιριάζουν όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά και με τις άλλες δηλώσεις Έχουμε μια συγκεκριμένη δήλωση όπως στην οποία θέλω να πιστήσω την προσοχή σας γιατί απαντά σε μια συγκεκριμένη ερώτηση που ετέθη αυτό το opt-out από την προσωρινή εφαρμογή. Αυτό δεν υπάρχει κάποια κρατημέλη θέλησαν να δηλώσουν ρητά κάποια πράγματα που απλά επαναλαμβάνουν την νομοθεσία που ισχύει για όλους. Αν σε κάποιο κράτος μέλος. Το όργανο το οποίο είναι επιφορτισμένο με την υπογραφή της συμφωνίας, ε, την οποία συμμετέχει το εν λόγω κράτος μέλος ως ε, ξεχωριστό είτε μονάδα είτε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν αυτό ακυρώνει τη συμφωνία, τότε αυτό το κράτος μέλος δεν μπορεί να την κυρώσει και αν είναι δική, δική της ε, συμφωνία, τότε πρέπει και να ενεργήσει ώστε να πάψει τη συνεφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας. Ε, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν μονομερώς να ε, πάψουν την εφαρμογή μιας διάταξης μονομερώς. Αν όμως δεν μπορούν να την υπογράψουν επειδή είναι αντισυνταγματική, τότε η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Θεσμό θα πρέπει να ενεργήσει ώστε να πάψει αυτή τη συμφωνία. Εκτός αν γίνει κάποια άλλη δράση ώστε να λήξει η αντισυνταγματικότητα. Η δεύτερη πτυχή αυτής της δήλωσης είναι ότι η αδυναμία κύρωσης μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα του αυτού που η δήλωση ορίζει άλλες συνταγματικές διαδικασίες που εξασφαλίζονται από το αριθμό της κύρωσης. Αυτή τη διατύπωση τη χρησιμοποιήσαμε κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους λόγω της, διαφορε... των... της των συνταγματικών διαδικασιών στα κράτη-μέλη. Σε αυτή την περίπτωση αυτό σημαίνει ότι, πώς να το πω δεν ξέρω, ότι τα κοινοβούλια είναι κυρίαρχα. Επίσης είναι κυρίαρχα και όταν αλλάζουν τη γνώμη τους. Δηλαδή ένα ψήφισμα ενό κοινοβουλίου μπορεί να είναι η τελευταία του λέξη, αλλά μπορεί και όχι. Και κανένα άλλο δεν το γνωρίζει εκτό από το ίδιο το κοινοβούλιο. Κανεί δεν μπορεί και να το ξέρει άλλο. Αυτό που λέει λοιπόν η δήλωση αυτή είναι ότι εάν μια από αυτές τις συνταγματικές διαδικασίες κοινοβουλευτική κύρωση, μία ή περισσοτερε καταλήξει σε μόνιμη και οριστική αποτυχία της διαδικασια κυρωση στο εν λόγω κράτος μέλος, τότε ξαναρχόμαστε στο ίδιο πρόβλημα ότι η συμφωνία αυτή δεν μπορεί να κυρωθεί και η προσωρινή τη εφαρμογή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να δράσει, να ενεργήσει. Τώρα, αυτό ισχύει όταν το κράτος μέλος θα κοινοποιήσει την οριστικότητα αυτής της απόφασης, τον οριστικό χαρακτήρα. Ε, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προδιαγραφή γι' αυτό και στα κράτη-μέλη δεν υπάρχει ήδη κάποια καθιερωμένη μορφή γιατί αυτά, τα πράγματα είναι αρκετά σπάνια. Ε, αυτό είναι το νόημα λοιπόν της δήλωσης το και αυτό που έχει σημασία επίση είναι η δήλωση του Συμβουλίου που απαντά στις δηλώσεις των κρατών μελών. Τα κρατημέλη ε, δηλώνουν κάποια πράγματα που είναι γενική εφαρμογή και το, το Συμβούλιο δηλώνει κάτι που είναι γενική εφαρμογή για τα ίδια τα κρατημέλη. Ακόμα δηλαδή και τα κρατημέλη που δεν έχουν συνδεθεί με τη δήλωση αυτή, εάν κοινοποιήσουν στην Ευρωπα... τα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι δεν μπορούν να κυρώσουν τη ΣΕΤΑ για οποιοδήποτε λόγο, είτε είναι θέμα ε, συνταγματικής συμβατότητας, είτε επειδή το Κοινοβούλιο δεν θέλησε να ακυρώσει και κατά την κρίση του εν λόγω κράτους μέλους αυτό είναι μόνιμο και οριστικό. Ε, τότε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να δράσουν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές ε, δραστηριότητες. Δυστυχώ, ειλικρινά πρέπει να σας πω, δεν ξέρω ακριβώ ποιε είναι αυτέ οι διαδικασίες. Το μήνυμο θα ήταν μια απόφαση του Συμβουλίου θα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο ή, να, ή απλώς να βάλουμε στο ράφι τη συμφωνία. Φαντάζομαι ότι αν πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο, μάλλον το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσουν την αρχική, την, ε, να ακυρώσουν αρχική ε, υπογραφή, επικύρωση. Θα το πρέπει να το δούμε αυτό, δεν ξέρω. Τώρα, αν είναι σοφό το ότι και μειχτό χαρακτήρα για αυτή τη συνθήκη ή όχι, ξέρετε τη θέση που έχει λάβει ο πρόεδρος Γιούνκερ δημοσία για αυτό το θέμα. Πάντως, όσον αφορά τούτο εδώ το κοινοβούλιο τώρα, με, ε, από νομική άποψη το, θέμα έχει κινηθεί. Το Συμβούλιο έχει λάβει απόφαση που είναι νομικό δεσμευτική να υπογράψει αυτή τη συμφωνία ως μεικτή συμφωνία. Τα κρατημέλη υπογράφουν χωριστά και η συμφωνία έχει διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο προς εξέταση και διαβούλευση. Τώρα, αν αυτό θα πρέπει να έχει γίνει διαφορετικά ή κάτι άλλο, δεν έχει τώρα νόημα ε, από νομικής άποψης. Το ίδιο θα ξαναπροκύψει στο μέλλον και θα έχουμε εντωμεταξύ λάβει κάποια διευκρίνηση από το 10. Μπορεί πολιτικός να είναι σκόπιμο μια τέτοια συζήτηση για τη ΣΕΤΑ, πάντως να σας διευκρινίσω ότι από νομικής άποψη δεν έχει πλέον νόημα. Ίσως να έχει νόημα για μελλοντικέ συμφωνίες. question of what happens uh, to provisional application during provisional application. During... Λοιπόν, τώρα για την ε, προσωρινή εφαρμογή θα αρχίσει η εφαρμογή και θα είναι επιχειρησιακά όλα, κοινή επιτροπή, όλα, μεικτή επιτροπή, ό,τι προβλέπετε. Κάτι που δεσμευτήκαμε να μην κάνουμε είναι να προτείνουμε στον Καναδά μια απόφαση της κοινή επιτροπής πριν να έχουμε την κρίση του ενός συνταγματικού δικαστηρίου που εξετάζει το συγκεκριμένο θέμα, το γερμανικό δηλαδή. Κάπου στο 17 θα βγει η απόφαση. Θα πρέπει να σας θυμίζω ότι σπάνια χρειάζονται αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής στις πρώτους μήνες προσωρινής εφαρμογής μιας συμφωνίας και αν κάτι προκύψει θα είναι διοικητικής φύσης. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι θα χρειάζεται να ενημερωθεί το όνομα κάποιων μονάδων στα παραρτήματα για τους ε, δημόσιες προμήθειες. Είναι πολλά διοικητικό θέμα, αλλά δεν είναι τόσο ουσιαστικό και μπορεί και να περιμένει. Επίσης αυτό είναι πολύ σημαντικό για το θέμα της, του προγράμματος εργασίας για το Διευθυντικό Δικαστήριο. Ε, εάν δούμε το ιστορικό των συστημάτων διατησίας και είχαμε τη συζήτηση αυτή επαναλημμένα σε αυτήν την Επιτροπή, το ICS θεωρήθηκε ως, ως θέμα υπό επεξεργασία και εξέλιξη. Αυτό που είχαμε προβλέψει για τη ΣΕΤΑ ε, το βλέπουμε αναθεωρημένο στο Συμφωνία για το Βιετνάμ και στη Συμφωνία για το Βιετνάμ βλέπουμε κάποιες ρήτρε για εισαγωγή κάποιων στοιχείων αμέσως μετά την έναρξη ισχύω. Στην περίπτωση του Καναδά αυτά τα στοιχεία ήταν λίγο πιο εκτεταμένα λόγω της ταχύτητας με την οποία έγινε η αναδρομική διόρθωση όταν έγινε. Τώρα, αυτό που η Βαλονία και μεταξύ άλλων, γιατί λάβαμε και παρόμοια αιτήματα από άλλα κράτη-μέλη ε, και ρωτούσε, ήταν ακριβώς η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Ήταν δηλαδή η δυσαφήνεια για την επιλογή των δικαστών. Ένα θέμα το οποίο το αφήσαμε αλήτω γιατί κάθε μέρος επιλέγει τους δικαστές όπως θέλει. Τώρα λέμε πώς θα διαλέξουμε εμείς τους Ευρωπαίους δικαστές και πώς θα παρακολουθούμε τις επιλογές των υπολείπων ε, δικαστών. Το θέμα του κώδικα διοντολογίας Έχουμε ηθικούς κανόνες τόσο στη ΣΕΤΑ όσο και στη Συμφωνία για το Βιετνάμ. Έχουμε πάρει διμερή δέσμευση να τα βελτιώσουμε όλα αυτά, να διευκρινίσουμε, να αποσαφηνίσουμε, να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Το μήνυμα από τη Βαλονία λοιπόν και από άλλους είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι διόριστο. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια. Ε, γρηγορότερα, αν δούμε αυτή τη δήλωση, λέει ένα πρόγραμμα, μάλλον ε, εκθέτει ένα πρόγραμμα εργασίας με βάση τους κανόνες της αρχικής ε, ε, πρότασης για το ICS και αυτό μέσω των ρητρών αναθεώρησης που υπήρχαν ήδη με τη συμφωνία. Αυτό που κάναμε είναι ότι αναλάβαμε μια δέσμευση να περιοδοτήσουμε τώρα αυτές τις ρήτες ε, αντί για αργότερα στο μέλλον και να πούμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε ώστε να επιτύχουμε αποτέλεσμα σε αυτήν την μεταρρύθμιση. Αυτό θα μπορούσε κανείς να το έχει μαντέψει και από τη συζήτηση που είχαμε ε, ήταν μια ε, περίπτωση χαρακτηριστική και εφόσον μπορούσε κανείς να το φανταστεί γιατί να μην το πούμε και να μην δεσμευτούμε. Και όλα ότι δεν θα αλλάξουμε τη γνώμη. Τώρα θα πρέπει να πείσουμε τον ε, Καναδά γιατί με ενθουσιασμό αγκάλιασε ο Καναδάς την, την ιδέα του ICS. Υπάρχει βέβαια πιθανότητα ο Καναδάς να μην συμφωνήσει και γι' αυτό και η Πολωνία και η Βελγική κυβέρνηση προστατεύθηκαν από αυτή τη δυνατότητα και είπαν ότι αν δεν γίνει αυτό δεν πρόκειται να ακυρώσουμε τη συμφωνία. Τώρα, πέρα από το γεγονός ότι και πάλι τα κοινοβούλια είναι κυρίαρχα και άμα σήμερα λένε ότι δεν θα κάνουμε το τάδε, αλλά αύριο αποφασίσουν θα κάνουν το τάδε, δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς γιατί είναι κυρίαρχα. Πάντως είναι ε, μια ισχυρή πολιτική δήλωση. Υπό ποιους όρους η Βαλονία θα δώσει την ε, έγκρισή της για την κύρωση της συμφωνίας. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι είναι σωστό έτσι κι αλλιώς. Πιστεύουμε πως ο Καναδάς θα συμφωνήσει πως είναι το σωστό και θα έχουμε το μέσο αυτό. Αυτό θα μας πάρει λίγο χρόνο. Ε, θα είναι λίγο περίπλοκο. Ε, μέχρι τότε θα έχουμε την απόφαση και του συνταγματικού, Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου και αν δεν το έχουμε θα μπορούμε να απελευθερωθούμε από την λήψη αποφάσεων από την Κοινή Επιτροπή και ε, θα μπορούμε αυτό να το εντάξουμε στη συμφωνία πριν, στη διάρκεια της προσωρινής ισχύς. Αυτό το είπαμε στη βελγική κυβέρνηση και στο Βαλλονικό Κοινοβούλιο, ότι δηλαδή είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Και η βελγική δήλωση που λέει πως ε, οι βελγικές ε, κυβερνήσει θα σχετίζονται με την εθνική του κυβέρνηση κτλ. Θα διευκρινίζουν και τι θα πρέπει να ε, κάνει ο καθένας. Πάντω, εμείς πιστεύουμε πως πρέπει να το κάνουμε αυτό και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εάν οποιοδήποτε ε, ευρωπαϊκός φορέας ε, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και τα Εθνικά Κοινοβούλια να παρακολουθούν τις ενέργειές μας. Για το θέμα του ΔΕΚ. Το ΔΕΚ ρωτήθηκε ποιες είναι οι αρμοδιότητες σε σχέση με τη Συμφωνία για τη Σιγκαπούρη. Να πω ότι η Συμφωνία της Σιγκαπούρης περιλαμβάνει ένα πρότυπο ISDS, δηλαδή διατησίες μεταξύ ιδιωτικού φορέα και κράτους. Και το σχέδιο συμφωνίας αναμένει την ανάπτυξη αυτής της συζήτησης και θα πρέπει να συνεχιστεί μετά. Όμως το δικαστήριο δεν μπορούσε να εξετάσει την αρμοδιότητα να κάνει κάτι για κάτι που είναι ασύμβατο με τη συνθήκη. Οπότε, εφόσον το δικαστήριο εξετάζει την ουσία του αιτήματος ε, για συμπεριλαμβανομένου του ποιος είναι ο αρμόδιος για το ISDS, τότε θα πρέπει να πιστεύει το, το δικαστήριο ότι το ISDS είναι συμβατό με τις συνθήκες. Δηλαδή, διαφορετικά θα είχε πει αυτό είναι σύμβατο με τις συνθήκες, δεν πρόκειται καν να το εξετάσουμε. Γιατί κανείς δεν έχει αρμοδιότητα να το κάνει. Βέλη, είχε τα έτοιμα της Βαλωνίας, αλλά επειδή και με τη συμφωνία άλλων ομοσπονδιακών ε, φορέων ε, δεν υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί το στο δικαστήριο να εκφράσει γνώμη για το ICS και τη συμβατότητα αυτού με τη συνθήκη. Δεν έχουμε καμία σκοπό, κανένα σκοπό να αναπτύξουμε ένα ICS το οποίο είναι ανασύμβατο με τη συνθήκη. Άρα λοιπόν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Τώρα, αν θα το κάνει το Βέλγιο, δεν το ξέρω. Είναι δικό τη κυρίαρχο δικαίωμα και κατά σύμπτωση το γεγονό ότι το Βέλγιο το έχει αυτό ξεκαθαρίσει δεν αλλάζει το γεγονό ότι οποιοδήποτε κράτο μέλο έχει την ίδια εξουσία και οποιαδήποτε θεσμικό ευρωπαϊκό όργανο μπορεί να κάνει το ίδιο. Και αυτή η απόφαση μπορεί να ληφθεί ανα πάσα στιγμή. Είναι δηλαδή μια φυσιολογική λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Ε, ήταν σημαντικό για το Βέλγιο να τονίσει, να δείξει πως σκοπεύει να το κάνει. Αλλά είναι κάτι το οποίο εμεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ως Κομισιόν. Αντίθετα, οποτεδήποτε υπάρχει γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπως έχουν τονίσει και κάποιοι βουλευτές εδώ, αυτό ενισχύει τη διαδικασία μας και δεν την αποδυναμώνει. Τώρα, λίγες λεπτομέρειες. Γεωργία. Υπενθυμίστηκε προηγουμένως και το επιβεβαιώνω ότι η ΣΕΤΑ δεν τροποποιεί την νομοθεσία μας για τα γεωργικά. Δεν τροποποιεί το γεγονός ότι δεν μπορείτε να πωλείτε κρέας με ορμόνες στην Ευρώπη. Δεν μπορείτε να ε, επεξεργαστείτε ζώα που έχουν τραφεί με ορμόνες στην Ευρώπη και δεν τα εισάγουμε ούτε από τον Καναδά ούτε από καμία άλλη πηγή είτε ε, ε, με, βάση δασμολόγιο ε, κάποιου διεθνούς οργανισμού ή όχι. Το ίδιο ισχύει, δηλαδή η ΣΕΤΑ δεν περιλαμβάνει διμερείς ρήτρες διαφύλαξης. Περιλαμβάνει η ΣΕΤΑ, μάλλον αφήνει άθικτα αθικτό το αμοιβαίο δικαίωμά μας Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τις διατάξεις του ΠΟΕ, αυτά δηλαδή που ισχύουν ήδη ως νομοθεσία. Η δήλωση που έχετε εκεί επαναλαμβάνει το γεγονό αυτό. Έχουμε την νομοθεσία αυτή και μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε εφόσον οι εισαγωγές από τον Καναδά πληρούν τις προϋποθέσεις. Το ίδιο για την πλευρά του Καναδά. Τώρα, εάν οι εισαγωγές υπό περιορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων μπαίνουν κάπου αλλού ή όχι, αυτό είναι διαφορετική ιστορία. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ απίθανο, διότι οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα πολύ υψηλά απαγορευτικά καθεστώτα εκτός ποσοστώσεων διασφαλίζουν συνήθως ότι θα μπει στόπι στις αγωγές πριν να προκριθεί η ε, επίκληση της ρήτρα. Υπάρχουν λοιπόν τα μέσα αυτά, τα εργαλεία αυτά και θα χρησιμοποιηθούν. Μίλησα για την ε, διαφύλαξη, την precaution. Ίσως πρέπει να πω λίγα λόγια για την ρυθμιστική συνεργασία. Και θα σταματήσω εκεί, Πρόεδρε. Η ρυθμιστική συνεργασία. Ένα θέμα που τίθεται συχνά και όχι για πρώτη φορά έχει ως εξής. Η ΣΕΤΑ δεν περιλαμβάνει υπερεθνικό όργανο που μπορεί να ρυθμίζει αυτό αντί της Ευρωπαϊκής Ενώσης ή του Καναδά. Εκτός από το γεγονός ότι υπάρχει ένας μηχανισμός στην ΣΕΤΑ για τη ρυθμιστική συνεργασία που είναι ωστόσο οικειοθελή, δεν επιβάλλει την συμμετοχή όπω λέει το instrument αυτό ακόμα και αν γίνει σε οικειοθελή βάση τα μέρη παραμένουν ελεύθερα να αγνοήσουν την έκβαση τη εφαρμογή του μηχανισμού. Και πέραν από αυτό, οτιδήποτε συμφωνήσουμε με τον Καναδά θα πρέπει να εφαρμοστεί μετά από απόφαση της Επιτροπής σας. Της Επιτροπής όπου συνεργάζονται τα δύο μέρη. Όπως και, όλες οι άλλες διεθνείς, και σε όλες τις άλλες διεθνείς συμφωνίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να ε, προβεί σε κάποια ενέργεια αν δεν έχει την εξουσιοδότηση. Διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κάτι το οποίο δεν έχει καμία ουσία. Η εξουσιοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το λιγότερο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο των Υπουργών. Συχνά θα πρέπει να είναι και η πλήρης διαδικασία με συνεργασία Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως αλλιώς δεν μπορεί να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διατάξεις του κεφαλαίου για την ε, ε, βιώσιμη ανάπτυξη είναι δεσμευτικές. Γιατί συχνά υπάρχει εδώ μια παρανόηση. Είναι απολύτως πλήρως δεσμευτικές και υπόκεινται σε ιδιαίτερο μηχανισμό και οι διατάξεις για τον ε, μηχανισμό ε, διαιτητικής επίλυσης επίσης είναι δεσμευτικές. Δεν μπορούν να πούν εάν διαφωνούμε με την απόφαση του Κοινοβουλίου δεν υπάρχει η απόφαση. Υπενθυμίζω την ομόφωνη θέση του Συμβουλίου και θέση την οποία έχει στηρίξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά επανάληψη ότι η χρήση εμπορικών κυρώσεων για την επιβολή ε, όρων στα εργασιακά και για την βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι δυνατή. Έχουμε μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η θέση αυτή μπορεί να αλλάξει. Όμω, για την ώρα η θέση που έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα τελευταία χρόνια είναι αυτή. Και δεν θα βρείτε τίποτε άλλο εκτό από αυτή την θέση. Αυτό που κάναμε για να ανταποκριθούμε μαζί με τον Καναδά στην ανησυχία αυτή είναι ότι θα προκαλέσουμε την επανεξέταση που προβλέπει η συμφωνία για να επανεξετάσει τη διάταξη αυτή μαζί και την δυνατότητα επιβολής, enforceability. Έχουμε δηλαδή το μηχανισμό για να φέρουμε την αλλαγή αυτή στην στη Συμφωνία με τον Καναδά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς που μας έδωσαν μερικά λεπτά παραπάνω. Έτσι ολοκληρώνεται το σημείο 22. Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους της Επιτροπής ότι έχουμε έφτακτη συνεδρίαση προβλέψη για, το, για την Σύνοδο του Στρασβούργου ώστε να επικεντρωθούμε μόνο στις νομικές πτυχές. Είπαμε όρο ότι θα γίνει και δήλωση της νομικής μας υπηρεσίας μόνο για το νομικό καθεστώς και κάποια θέματα σχετικά με το νομοθέτημα και την ε, δήλωση ή τις δηλώσεις καλύτερα. Μόνο για αυτό το θέμα έκτακτη συνεδρία στο Στρασβούργο. Μετά έχουμε ανταλλαγή απόψεων 29 Νοεμβρίου και κατάρτιση της έκθεσης από τον εισηγητή. Και ανταλλαγή απόψεων και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Στο 24 τώρα σας ρωτώ αν υπάρχει κάτι άλλο, στα διάφορα όχι. Προσεχή συνεδρία 28-29 Νοεμβρίου και σας ευχαριστώ.